Is it possible to start? Hello? Should we start? Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ουρασία διάταξη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ανακοινώσει Προέδρου. Ω συνήθω να σας πω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση, στο e-meeting και υπάρχει και το ενημερωτικό δελτίο. Θα θυμάστε ίσως ότι στην τελευταία μας συνεδρίαση είχα ε, πει ότι οι κατάληψη ψηφοφοριών θα διατίθενται ηλεκτρονικά πλέον. Βέβαια, λάβαμε πολύ σύντομα μετά από αυτή την ε, συνεδρίαση ένα πολύ ευγενικό email ενό δημοσιογράφου που προσπαθεί να παρακολουθεί προσεκτικά τις εργασίες του Κοινοβουλίου και μα είπε πόσο του βοηθούσε να μπορούν να παρακολουθούν του καταλόγου ψηφοφοριών και πόσο πολύ τους βοήθησε σε σχέση με άλλες επιτροπές που δεν το κάνουν, ιδίως στην ΕΚΟΝ. Είπα ΕΚΟΝ, ο... Τέλος πάντων. Να ευχαριστήσω λοιπόν πολύ τη γραμματεία που αναρτά στο διαδίκτυο και τις, κατα, τους καταλόγους ψηφοφοριών και ελπίζω να μιμηθούν το παράδειγμά μας και άλλες επιτροπές. Θα το συζητήσω με τον ε, αξιαγάπητο κύριο Γκουαλτιέρη συντόμους. ενημέρωση μάλλον σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους και διάφορες διοργανώσεις. Να μιλήσω για τον τριμερή διάλογο για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μία πρώτη συνεδρίαση για τον τριμερή διάλογο για την ενιαία αγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Θα θυμάστε ότι ψηφίσαμε το κείμενο του Κοινοβουλίου πριν από περίπου ένα χρόνο και χρειάστηκαν σχεδόν 12 μήνες για να καθίσουν ε, στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων ε, οι τρεις πλευρές. Είχαμε λοιπόν ε, μακροσκελής ανταλλαγής απόψεων για τα βασικά ζητήματα. Βέβαια, εισηγητής είναι από την Επιτροπή Ήτρε, συγκεκριμένα η Πιλάρ Δελκαστίγιο. Στόχος είναι να γίνουν σεβαστές θέσεις του Κοινοβουλίου, ιδίως ό,τι αφορά την κατάρρευση του roaming, της περιαγωγής και την ανάγκη να έχουμε μια αποφασιστική προσέγγιση υπέρ της ουδετερότητας ε, του διαδικτύου. Υπήρχαν πολλές παρεμβάσεις και από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξέφραζε τη λύπη για το ότι δεν αναφέρεται τίποτα για το θέμα του φάσματος στο κείμενο του Συμβουλίου. Το φάσμα όμως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αν θέλουμε οι υποδομές ψηφιακές να είναι καλύτερες στην Ευρώπη. Συνολικά και εγώ επίσης πολλές φορές έλαβα το λόγο και μίλησα για την τελική χρήση και τα δικαιώματα, τα δικαιώματα μάλλον των τελικών χρηστών. Και ελπίζω να αναφέρονται πολύ περισσότερα για την διαφάνεια και την ενημέρωση των καταναλωτών, πάντως στο πλαίσιο των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. Να είναι δηλαδή αυτές οι διατάξεις το επόμενο, στην επόμενη δοχή του κειμένου. Το Συμβούλιο είπε ότι θα το ξαναμελετήσει. ιδίως τα περί ενημέρωση των ε, τελικών χρηστών, συμβόλαια, ε, πρόορη ε, διακοπή της σύμβασης εφόσον δεν παρέχει αυτά τα οποία είχε προβλεφθεί να παρέχει η σύμβαση κτλ. κτλ. Αν θέλουμε να έχουμε μια νέα αγορά τηλεπικοινωνιών πρέπει να είναι συγκρίσιμα τα συμβόλαια και συμβάσεις να μην γνωρίζουν μόνο τις χρεώσεις παραδείγματος τη περιαγωγή, αλλά να έχουν στοιχεία για τα συμβόλαια. Ελπίζω λοιπόν να συμπεριληφθούν ε, τέτοιε διατάξει στο κείμενο. Βέβαια η Λεπτονική Προεδρία ξεκαθάρισε ότι εάν θέλουμε να έχουμε διαπραγμάτευση ε, μιας δέσμης μέτρων για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών στη δική του Προεδρία, δεν μπορούν να βάλουν μέσα εκεί ένα κεφάλαιο για το φάσμα. Γιατί δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο, είπαν. Γι' αυτό και εστιάζουν στην ουδετερότητα του διδεκτήου και την περιαγωγή. Αλλά δεν μπορούν επί λεπτονικής προεδρίας ε, να κάνουν ε, περισσότερη δουλειά πάνω στο θέμα του φάσματος. Αναμένεται επόμενο τριμερή διάλογο σε κάποιε εβδομάδε. Θα συνεδριάσουμε και στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων. Θα σα ενημερώσω όποτε έχω κάτι νεότερο. Για τη δική μου τώρα πολιτική ομάδα ήμουν μόνιμη συγγήτρια από την Επιτροπή Ήτρε, για την Επιτροπή Ήτρε, από την πολιτική μου ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος από την ομάδα ECR να με αντικαταστήσει. Εγώ, επειδή είμαι εισηγήτρια για την εσωτερική αγορά, θα εμείνω σε αυτά δεν ξέρω αν θέλετε να διαχωρίσω τις δύο ιδιότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίθετη πρόταση. Ξέρετε ότι θα συνεχίσω να προασπίζω τις ε, θέσεις της δικής μας Επιτροπής. Έρχονται και άλλοι σιγά σιγά, οπότε τώρα μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε στην γνωμοδότηση της Μαρλέν Μίτσι για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εξέταση των τροπολογιών. 244 τον αριθμό. Να δώσω το λόγο ευθύς αμέσω στην εισηγήτρια, την οποία και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, τεράστιος αριθμός των τροπολογιών. 113 κατέθεσα εγώ και 131 κατέθεσαν οι ομάδες S&D, EPP, CR, GUE, η μη εγγεγραμμένη, σχεδόν όλες τις πολιτικές ομάδες δηλαδή. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα και ότι υπάρχει απόκληση αλλά και σύγκληση απόψεων. Στόχος μας βέβαια είναι να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα, να αυξήσουμε την απασχόληση, να συμβάλλουμε στην ε, οικονομική ευρωστία ουσιαστικά. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσης αυτής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς έχουμε τους ίδιους στόχους, αλλά με διαφορετικούς ε, τρόπους από αυτούς προτείνονται. Είναι πάρα πολλέ τροπολογίε, άρα θα περιστώ στι σημαντικότερε. Δεν μπορώ να τι καλύψω όλε. Ξεκινά λοιπόν με την 116 τροπολογία από διάφορα μέλη της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, της ΙΜΚΟ και των Επιτροπών Γιούρι και Έμπλη, έχει κατατεθεί αυτή τροπολογία. Και ζητεί τελικά την ε, απόρριψη της όλης πρότασης της Κομισιόν. Αυτή είναι και η γενική γραμμή της δικής μου πολιτικής ομάδας, οφείλω να σας πω. Τούτου λεχθέντος, ένα άλλο επίμαχο σημείο, ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε ακριβώς εκεί. Υπάρχει απόκληση απόψεων. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 21 το καθεστώς Πρέπει να διαγραφεί αυτό και οι σχετικές τροπολογίες. Υπάρχουν επίσης αρκετές τροπολογίες οι οποίες ε, ασχολούνται με το κατά πόσον θα πρέπει να επηρεαστεί και η εθνική νομοθεσία. Υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει αυτό. Άλλο είναι το έβρος αυτής της νομοδότησης και πολλές τροπολογίες συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ρυθμίσεις περί εταιρικού, ο νόμος εταιριών δηλαδή της κάθε χώρας. Πλήρης εναρμόνιση των εθνικών ε, νόμων δεν είναι κάτι απαραίτητο, δεν είναι ένα στόχος και συμφωνώ και εγώ. Ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι η νέα έδρα και εδώ έχουμε αρκετές τροπολογίες. Η ιδέα είναι ότι το φορολογικό δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο της χώρας καταχώρησης, της ώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση πρέπει να είναι αυτό που θα ισχύει. Εδώ πιστεύω ότι υπήρξε αρκετή σύμπνοια. Σε ό,τι αφορά το καταστατικό, ήταν και αυτό ε, ένα ζήτημα που με το οποίο ασχολούνται πολλές ε, τροπολογίες, τι πρέπει να περιλαμβάνει. Έχουμε την τροπολογία 103 Άντερσον Κοφεράτη, είναι καλή τροπολογία γιατί προτείνει μια λύση στο πρόβλημα της ε, ιωνία Έχουμε θέματα επίσης με την επιγραμμική καταχώρηση και την αναγνώριση, το identification, πώς θα είναι ε, βέβαιο ότι πρόκειται για αυτά τα άτομα τα οποία εγγράφονται στο διαδίκτυο. Επίσης έχουμε το κεφαλαίο και τη... τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Το μετοχικό κεφάλαιο νομικά αποθεματικά είναι ένα θέμα, αν πρέπει να έχουμε τέτοια αποθεματικά και σε τι πρέπει να συνίστανται αυτά. Αυτά είναι τα επίμαχα σημεία τα σημεία τριβής. Νομίζω όμως ότι σίγουρα πρέπει να έχουμε απλούστευση, μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας και πιο πολλές επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν, να μπουν σε αυτή την ενιαία αγορά. Αυτό που δεν πρέπει όμως να κάνουμε είναι να θυσιάσουμε την ε, ποιότητα σε βάρος της, ή μάλλον υπέρ της ποσότητας. Όλοι θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα επίπεδο καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ελπίζω πάντως να καταφέρω να συμβιβάσω τις διάφορες ε, αποκλίνουσες απόψεις. Sorry. Um, for the EPP, Stefan, Ivan Stefanis. Ivan Stefanis από το ΕΛΚ. Και Madam Chair. Ευχαριστώ Γενικά υποστηρίζω την πρόταση αυτή που προετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι πρέπει τον στόχο αυτή της ε, πρότασης να τον διατηρήσουμε, δηλαδή να μπορούν να καταχωρούν ευρύτατα και χωρίς δαπάνες οι εταιρείε αυτές για να λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. Να είναι λοιπόν, ας το πω έτσι, η δυνατότητα χαμηλού κεφαλαίου το πολύ πολύ ένα ευρώ ώστε να μπορεί διαδικτυακά να καταχωρείται κανείς. Και θα πρέπει λοιπόν έτσι το γραφειοκρατικό κόστος να μειωθεί οπωσδήποτε. Κατανοώ τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και επιφυλάξεις και εδώ βρισκόμαστε για να αναζητήσουμε συμβιβαστικές λύσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαπίστευση, για παράδειγμα, που θα πρέπει να γίνεται στα κράτη-μέλη. Και είναι δουλειά των κρατών μελών να δουν ποια συνέχεια θα δίνεται αν θα διατηρηθούν οι φυστάμενες διατάξεις ή αν θα, θα τροποποιηθούν. Επίσης για ένα συμβασμό που προσπάθησαμε να βρούμε για τις ε, νομικές πτυχές. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε το βασικό μας στόχο έχοντας υπόψη να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και να μειωθεί η δαπάνη η οποία θα συνεπάγεται, την οποία θα συνεπάγεται αυτό ώστε νέοι επιχειρηματίες να βοηθηθούν διότι τους χρειαζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη. Μια και η απασχόληση είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητα της Ευρώπης σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ και εμείς από την ECR συμφωνώ εγώ με την πρόταση που έγινε Υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η καλύτερη οδός να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες που προσυπογράφονται και από άλλα μέλη και με την υποστήριξη του κ. Γκούγκερ για την βελτίωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως διατηρώντας τα ουσιώδη στοιχεία τα οποία ζητεί να υπάρξουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν συμφωνούμε με την, στο σχέδιο γνωμοδότησης για την ε, αναζήτηση με μια νέα μορφή που θα περιορίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επικεντρώνω τις τοπολογίες μου σε αρκετά κέρια σημεία. Έχουμε όμως ε, την άποψη ότι σε κάποια σημεία πρέπει η εθνική νομοθεσία να λειτουργήσει και έχουμε μια ανοιχτή προσέγγιση υπέρ των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να παραμείνουν στην αμοδιότητα των κρατών μελών και ευρύτερες αποφάσεις να μπορούν από την επιμέρους εταιρεία να λαμβάνονται. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεσπίσει τα κριτήρια για αυτές τις επιχειρήσεις. Οι καθημερινές απαιτήσει λειτουργίας όμως θα πρέπει να είναι υπόθεση άλλων φορέων των εθνικών νομοθετών. Πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ηλεκτρονική, διαδικτυακή δηλαδή καταχώρηση για παράδειγμα και απαιτήσει κεφαλαίου που είναι ένα κύριο σημείο αυτού του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι το δυνατόν μικρότερες αυτές οι απαιτήσει. Δηλαδή να υπάρξουν οι λιγότεροι περιορισμοί σε σχέση με την ίδρυση επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει απλά και μόνο να βρίσκονται κάποια χρήματα για να διεκπαιρεωθεί μια γραφειοκρατική διαδικασία και μόνο. Είμαστε υπέρ του ότι οι απαιτήσει κεφαλαίου πρέπει να είναι στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Ένα ευρώ παράδειγμα. Η άλλη παρατήρησή μου αφορά την πρόθεση και ως νομοθέτες δεν πρέπει να φοβόμαστε να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να αποτύχουν. Πολλές φορές ε, προέρχονται εταιρείε, ε, επιχειρήσεις από εταιρείε ή επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποτύχει κατά το παρελθόν. Εφόσον λοιπόν όσο αφορά την πτώχευση ή τη χρεοκοπία υπάρχουν ρυθμίσεις ε, που διέπουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να φοβόμαστε να αφήσουμε εταιρείε να αποτύχουν. Οι πολιτικές στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι κυρίως ενθαρρυντικές ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να δραχθούν τις ευκαιρίες να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Και με αυτό το πνεύμα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Tony G. Thank you. That's much easier to call me that Ευχαριστώ. Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να σχολιάσει κανείς. Μου αρέσει. Λοιπόν, θα έλεγα αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Να θυμόμαστε ότι οι νέοι βρίσκονται διασυνδεδεμένοι και πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται με αυτούς. Υπάρχουν προβλήματα, η καταχώρηση διαδικτυακά θα πρέπει να είναι καινούρια, νοπή εμπειρία. Μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη αυτή η διαδικασία Πρέπει να δώσουμε σκληρή μάχη, να είναι εύκολες και ε, ε, χωρίς γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις οι διαδικασίες. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ένα νομικό καθεστώς που επιτρέπει οι πολίτες να ψηφίζουν διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Λοιπόν, η ίδρυση εταιρεία και η λειτουργία εταιρεία διαδικτυακά, ηλεκτρονικά πρέπει να μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει να είμαστε προσεκτικοί, μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου κάποια κράτη-μέλη θα δίνουν ε, μάχη για να έχουν κάποιες ε, ε, εξουσίες για να πηγαίνουν στο σπίτι κάποιου για να καταχωρείται μια εταιρεία. Η όλη ιδέα είναι να είναι ένα απλό πλαίσιο αυτό το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει για αυτές τις εταιρείες. Να μην επιβαρυνθούν οι διαδικασίες γραφειοκρατικά. Πρέπει να παραμείνουν απλές και εύκολες και η ψηφιοποίηση. Όλα αυτά πρέπει να είναι ψηφιακά. Αυτό είναι το κλειδί. Πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει χαμηλότερη γραφειοκρατική επιβάρηση, μικρότερη γραφειοκρατική επιβάρηση. Μπορούν οι υποχρεώσεις μιας εταιρείας και οι συναλλαγές της να διεκπεραιώνονται ψηφιακά. Και ένα ευρώ είναι αρκετό <laughs> κεφάλαιο για να ξεκινήσει κανείς έτσι και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δράση ως αρρωγός της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ε, δηλαδή να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν ε, μια χορηγία, μια υποτροφία, μια χορηγία για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τους νέους να ε, δημιουργήσουν εταιρείες θα ε, είναι πραγματικά ενθουσιώδης, Θα δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους βοηθήσει και θα έχουν μια ευκαιρία να δράσουν. Και αυτό μπορεί να είναι μια επανάσταση, μια επαναστατική τροπή. Είναι πολύ μικρό το ποσό για το σύνολο του προπολογισμού, όμω δημιουργεί πολλέ θέσει απασχόλησης. Για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, κάτι κάνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ενθουσιώδει, με πάθος να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Μαστάκα. Um, συγγνώμη. Και ε, για τους πρασίνους θα, θέλατε, να, θα ήθελε ο εκπρόσωπος να λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, περιμένω να βάλω τα ακουστικά σας. Θα προσπαθήσω να τα πω καθαρά και εξάστερα και με ηρεμία αφού οι δημοσιογράφοι τόσο χαίρονται που μπορούν να μας παρακολουθούν ηλεκτρονικά. Καταρχάς, να ότι η Ζούλια Ρέντα δεν μπορούσε να έρθει. Οι πράσινοι βέβαια ε, στηρίζουν, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα μόνο και γι' αυτό δεν μπόρεσε να εκφραστεί σε σχέση με αυτή την τροπολογία. Όμως ε, συμφωνούν οι πράσινοι να διαβάσω λοιπόν αυτά που μου ζήτησαν να διαβάσω η Τζούλια. Η πράσινη λοιπόν είναι μεν επιφυλακτική απέναντι αυτή την πρόταση και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εντοπίζουμε όχι τόσο την αξία όσο του κινδύνου. Εμεί θέλουμε να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό ιστό. Υπάρχει όμω μεγάλο περιθώριο καταχρήσεων. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων εταιριών γραμματοκιβωτιών που χρησιμοποιούν μεγάλη όμιλη για να μην πληρώνουν του φόρου του. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι προκύπτουν ερωτηματικά με αυτή την πρόταση, που θα μπορούσε να βλάψει και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ποτέ ουσιαστικά δεν βρίσκουν ή δεν ξέρουν ποιο είναι ο ιδιοκτήτη μια εταιρεία, ο υπεύθυνο δηλαδή, και όλα αυτά πλήττουν και τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Θα παρακολύσει και τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων μια τέτοια πρόταση, κάτι όμω που είναι σημαντικό στην αγορά αυτή. Για όλους αυτούς τους λόγους η ομάδα των Πρασίνων θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να απορριφθεί αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Thank you. And Yuri has just arrived. Κύριος Μαστάλκα έφτασε. In which case, Andreas Schwab. Στην περιπτωσία ο κύριος Schwab. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση. Νομίζω ότι σε αυτή την Επιτροπή υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία ε, να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι πολίτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα να μπορούν να το κάνουν αυτό πολύ γρήγορα και όλες οι γραφειοκρατικές δυσκολίες ε, να ξαφανίζονται. Θεωρούμε λοιπόν ότι όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα φαινός και την ανάληψη ευθυνών Λοιπόν, ε, κατά την είδηση τη αφετέρου. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε με μία μόνο λέξη ότι είμαστε κατά της ε, γραφειοκρατίας. Βεβαίως ε, και όσον αφορά την ίδρυση εταιρεία υπάρχουν πολλά θέματα τα, πρέπει, τα οποία πρέπει να πλουστευτούν περαιτέρω. Βεβαίως και υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Εγώ όμως νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η ίδρυση μιας εταιρείας να μην ε, ε, καταλήγει σε φούσκα ε, γιατί κανείς τελικά υπάρχει κίνδυνος να μην γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνο για την ίδρυση αυτής της εταιρείας. Εγώ λοιπόν θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν λόγω αυτών θα μπορούσαμε να καταγράφουμε τις επιχειρήσεις ε, και ε, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άρα δηλαδή αυτός είναι ένας βατός δρόμος, εξαλείφθη τις δυσκολίες και θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Η κυρία Γκέπχατ και μετά η Μαρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο που έκανε πολύ καλή και σκληρή δουλειά μέχρι σήμερα και δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση αυτό το πράγμα, διότι μια απλούστευση των ε, επιχειρήσεων ωραίο πράγμα είναι αλλά και εγώ πιστεύω ότι η απορρίθμιση δεν είναι υποχρεωτικά πάντα η σωστή απάντηση και σε αυτούς τους τομείς και ιδιαίτερα σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπάρχουν πάρα πάρα πολλές οπές, πολλές χαραμάδες για να μπορεί να διαφύγει κανείς. Ιδιαίτερα όσον αφορά και τα δικαιώματα εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Πρέπει αυτές οι οπές, αυτές οι τρύπες να κλειστούν. Να μην μπορεί κανείς να διαφύγει. Πολλά πρέπει να γίνουν σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούμε να πούμε θα κάνουμε μια απορρίθμιση τελεία και παύλα. <clears throat> Οι μεγάλες επιχειρήσεις <clears throat> σε σχέση με τις ε, εταιρείε αυτές θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν για παράδειγμα να έχουν μια διαλειτουργία και να λειτουργήσουν σε άλλη χώρα πρέπει να μεριμνήσουμε πολύ προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτού του είδους οι μονοπρόσωπες εταιρείε θα διαμορφωθούν να συζητηθεί σε βάθος και εγώ έχω δυσκολίες με την απλή καταχώρηση ηλεκτρονικά διαδικτυακά Πρέπει και εδώ να μεριμνήσουμε πραγματικά να διασφαλίζεται επιτέλους ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση τέτοιου είδους καταχωρήσεων. Να μην υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δυνατότητες και ένα σύστημα πιστοποίησης ε, να βρίσκεται πίσω από αυτό την λειτουργία τα άτομα τα οποία θα ιδρύουν τέτοιες επιχειρήσεις να είναι πράγματι τα, τα άτομα που θα είναι οι μέτοχοι των εταιριών αυτών. Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να ρυθμιστεί. Πρέπει σε βάθος να προβληματιστούμε, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ όμως παρόλα αυτά και πάλι για την πολύ καλή δουλειά. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στη συντάκτρια αλλά και σε όλους τους κοιόδης εισηγητές. Πολλές τροπολογίες κατατέθηκαν και βλέπουμε ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμφέρον να προσπαθήσουν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταλήξουμε σε μια λειτουργική πρόταση που θα βοηθά τις επιχειρήσεις και δεν θα δημιουργεί προβλήματα. Συμφωνώ με τον Ανδρέα Σβάμπ να μην υπάρξει μια φούσκα μακροπρόθεσμα όσον αφορά την οικονομία. Δεν επιτρέπεται μόνο βραχυπρόθεσμα θέματα να αντιμετωπίζουμε πολλές επιχειρήσεις ε, θα καταχωρηθούν λέγεται και θα υπάρξει θετική εξέλιξη, θετική απήχηση. Όμως μακροπρόθεσμα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Επιχειρήσεις μπορεί καμιά φορά να χρεοκοπήσουν ή να πτωχεύσουν και μέσω της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλες επιχειρήσεις ε, μπορεί να ε, αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και πρέπει να δούμε για την καταχώρηση πώς θα λειτουργούν τα πράγματα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά με αθέμητο ανταγωνισμό. Οι μονοπρόσωπες εταιρείε λοιπόν μπορεί να μην είναι εκείνες οι οποίε ε, μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνε. όμως υπάρχουν ε, άλλες πτυχές για την εταιρική ευθύνη και τι υποχρεώσει υποχρεώσεις αντιμετώπισης τους των ευθυνών αυτών. Δεν πρόκειται μόνο για κάποιες εταιρείες ε, εικονικές ε, που έχουν απλά μια διεύθυνση, ε, ένα γραμματοκιβώτιο, μια εικονική διεύθυνση. Μπορεί για παράδειγμα στο όνομά μου να ζητηθεί να ιδρυθεί μια μονοπρόσωπη εταιρεία. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται το ότι έχει κανείς την έδρα του και κατοικεί στον ε, ε, τόπο ε, καταχώρησης της εταιρείας αυτής. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις ευθύνες των υπεύθυνων αυτών των εταιριών να τις ρυθμίσουμε με τρόπο που θα είναι λειτουργικός. Στις δικές μου τροπολογίες τι αναφέρω, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα έχουν ευθύνες και θα είναι υπεύθυνοι, θα μπορούν να λογοδοτούν οι ε, επικεφαλείς ε, διευθυντές. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων μία που θα λειτουργεί, μια κατηγορία που θα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο ευθυνών για τους α, ε, ε, διευθύνοντες και μια άλλη κατηγορία εταιριών όπου δεν θα υπάρχουν τέτοιες ευθύνες. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνεται αυτή η καταχώρηση και από ποιον. Έτσι λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει δεν μπορεί να εγκριθεί, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Thank you very much. Um, everybody's contribution was... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσα είπατε ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και προφανώς πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά κατά νου όσον αφορά το σχέδιο της εγγραμματοδότησης. Αυτά που είπε η Μαρία μόλις είναι πολύ σημαντικά. Ε, για να σεβαστούμε λοιπόν το εταιρικό δίκαιο και το εργατικό δίκαιο ενός μέλους πρέπει να γίνει αυτή η διαγραφή που αναφέρθηκε. Άρα δηλαδή ό,τι ισχύει τώρα στα κράτη-μέλη τώρα, θα ισχύει και για την ηλεκτρονική καταγραφή των εταιριών. Αυτό ήθελα να πω ε, και θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις για τη συνεισφορά τους και ελπίζω να εξευρεθεί κάποια λύση, τουλάχιστον ε, είμαι αισιόδοξη και εμείς ευχαριστούμε για τη δουλειά σας, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε. Ευχαριστούμε όλους ε, για τις παρεμβάσεις τους. Στις 23 Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στις 7 Μαΐου. Και θέλω να προχωρήσουμε το δυνατών στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα. Ε, για την έκθεση Κάθριν Στάιλον σχετικά με την νέα συνένεση για την εφαρμογή ε, των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι η έκθεση της Κάθριν ε, Στάιλον για την έκθεση που συντάχθηκε από την Νομική Επιτροπή. Συμβαστική πρόταση Ένα υπέρ κατά εγκρίνεται. Η υπέρ κατά εγκρίνεται η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ συγγνώμη η συμβαστική 3 είναι σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11, ε, 11 υπέρ κατά αποχές. Ε, μισό λεπτό, εδώ θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Την 11. Έκλεισε ο κατάλογος, εγκρίνεται. Η 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14, 15 μέχρι 19 κατέπεσαν. Καλύπτονται από τη συμβαστική πρόταση. Πάμε στην 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ κατά τα αποχές εγκρίνεται η 30 με την προφορική τροπολογία ε, της κυρίας Ρίντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 31 υπέρ κατά αποχές ε, καταπίπτει η 32 καταπίπτει η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 34 αποσύρθηκε η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 37 ε, διαγραφή υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε συνολικά για το σχέδιο της γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. εγκρίθηκε 33 υπέρ ένας ε, κατά τρεις αποχές συγχαρητήρια. Για όσους ήρθαν από άλλες επιτροπές προσπάθησα να τηρήσω το χρόνο. Τώρα, ε, σας καλωσορίσαμε, σας καλωσορίζουμε μάλλον. Τώρα πάμε στη δεύτερη έκθεση που είναι επίσης γνωμοδότηση από την Κάθιν Στάιλα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Τώρα, ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 με προφορική τροπολογία τη ε, της Βεζινή Ροζιέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Είναι η 14 για την οποία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Καταπίπτει ε, απορρίπτεται αν θέλετε, συμβαστική 3, το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ε, παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος, για το πρώτο τμήμα της συμβαστικής πρότασης 3. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής πρότασης 3, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 21, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4 συμβαστική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 29, παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει, παρακαλώ. Εγκρίνεται. Αυτή ήταν η 29. Η συμβιβαστική 5, το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται. Να το ξαναελέγξουμε παρακαλώ. και η 5 για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ ε, κατά αποχές ε, και η 39 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, ε, ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική έξι παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 με προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ κατά αποχές. Νομίζω αυτή απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Είναι η 53. Ε, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην παράγραφο 54. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 11. Παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η τροπολογία 63 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Γιατί η συμβαστική 9 το δεύτερο τμήμα. εγκρίνεται με μία ψήφο συμβιβαστική ε, 9 τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 70 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η σημαστική 10, το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ε, ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της συμβαστική 10. Απορρίπτεται για μία ψήφο και τέσσερις αποχές. Πάμε τώρα... Μισό λεπτό. Αυτή ήταν η 72 που απορρίφθηκε. Είπαμε η συμβαστική 10 την ολοκληρώσαμε και φτάνουμε στο τέλος ε, του καταλόγου ψηφοφοριών, ε, αυτής του καταλόγου ψήφου και ε, ψηφίζουμε για το σύνολο της έκθεσης ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε λοιπόν με 34 και 3 και 2 εποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτό το σημαντικό μέρος της εργασίας σας. Προχωράμε στη γνωμοδότηση τώρα για τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις για την διατλαντική Συμφωνία Επενδύσεων και Συναλλαγών TTIP ε, για την Επιτροπή μας είσαστε εσείς. Νομίζω έχετε την πρόθεση να παρέμβετε. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επικαιροποιήσω τους συναδέφους. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΠΑ υιοθέτησαν την κοινή δήλωση για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες που ευθυγραμμίζεται με το δικό μας συμβιβαστικό κείμενο και λέγεται ότι θα εξαιρούνται οι δημόσιες αυτές οι υπηρεσίες από τις ε, διαπραγματεύσεις της συμφωνίας. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν ανησυχίες των πολιτών και να μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε σε άλλα σημαντικά θέματα αυτών των διαπραγματεύσεων. Για τη δική μας γνωμοδότηση θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την συνεργασία τους. Συμβιβασμοί που θα ψηφιστούν προσυπογράφονται από συντριπτική πλειοψηφία κοινοβουλευτικών ομάδων για θέματα μεγάλης σημασίας για την δική μας Επιτροπή. Αυτά είναι τα κύρια μηνύματα που επιθυμούμε να αποστείλουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και όσον αφορά και τις δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες ε, ε, αγορές, προμήθειες ε, κτλ απογοητεύτηκα από το τελευταίο συμβαστικό κείμενο για το ISDS, διότι θεωρώ ότι αυτό δεν βρίσκεται στις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν να παραμείνουμε στην μεγάλη εικόνα των ζητημάτων αυτού του θέματος όπως ε, περιέχονται και ψηφίζοντας να το λάβουμε αυτό υπόψη. Δεν μπορώ να δώσω τον λόγο να παρέμβουν άλλοι σε αυτή τη φάση, εκτός αν είναι απόλυτα αναγκαίο και έχει κάποια σχέση με τον πίνακα για την ψηφοφορία που έχουμε ε, μπροστά μας. Θα υπάρξουν ούτως ή άλλως ανταλλαγές απόψεων επ' αυτών των θεμάτων. Προπολογίες 1 και 2 οι 3 και 4 πάνε από κοινού υπέρ, κατά. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την 3 και την 4 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Κατά τροπολογίες ισοψηφία, οπότε αρνητικό το αποτέλεσμα. Ε, συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 47 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 22 υπέρ κατά αποχές Καταπίπτει, το συγγνώμη, 22 καταπίπτει. Τώρα λοιπόν πάμε στην 21. Υπέρ, παρακαλώ, της 21, κατά, απόχες, απορρίφθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 49 αποσύρθηκε. Η 50 τώρα υπέρ, κατά, αποχές ε, καταπίπτει 51 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 203 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 220 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 205 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 157. Θέλει κάποιος να ζητήσει κάποιο έλεγχο. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε θα μπορέσουμε να ελέγξουμε σε σχέση με την διαμόρφωση πλειοψηφίων. 157 τώρα λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. πίπτη. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. πίπτη. 53 υπέρ. Κατά αποχές καταπίπτει 54 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 57 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 59 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 60 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβαστική τροπολογία 3 τώρα υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συγγνώμη εγκρίθηκε εγκρίθηκε η συμβαστική τροπολογία 3 εγκρίθηκε φυσικά τροπολογία 65 τώρα υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 70, τεχνικής φύσεως τροπολογία. Η 71 τώρα, υπέρ, κατά, άποχες, καταπίπτει. Η τροπολογία 20, υπέρ, κατά, άποχες, καταπίπτει. Η τροπολογία 75, υπέρ, κατά, άποχες, καταπίπτει. 77, υπέρ, κατά, αποχές καταπίπτει 79 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 72 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει και 94 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει πάμε στην 74 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 115 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 81 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 95 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 83 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 85 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβαστική τροπολογία 5 με προφορική τροποποίηση του ΕΛΚ όσοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 88 ως προσθήκη στη συμβαστική τροπολογία 5 Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Καταπίπτει. Η συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Καταπίπτει. Συγγνώμη, τι λέω. Μάλιστα. Εγκρίθηκε. Σωστό. Εγκρίθηκε η συμβαστική 6. Προσπαθώ με βραδύ ρυθμό να προχωρήσουμε ώστε αν χρειαστεί να μπορέσουμε να κάνουμε έλεγχο. Οποιοςδήποτε το ζητήσει θα γίνει αμέσως έλεγχος. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 110 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ε, τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 118 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 122 υπέρ η 122 λοιπόν υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο. Είναι τεχνική φύση η άλλη τροπολογία. Η 8 υπέρ συμβαστική τροπολογία κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην 149 τροπολογία υπέρ. Όχι, ναι, ναι, 149. Νέα παράγραφος, 7α δηλαδή, υπέρ της 149, κατά αποχές καταπίπτει 147 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 150 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 152 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η τροπολογία 155, που είναι προσθήκη στη συμβαστική 9, συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ της 155, κατά, αποχές, καταπίπτει. Τροπολογία 161, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 165, υπέρ, όχι, όχι, λυπούμε. Εντάξει, αυτή καταπίπτει. Δεν θα ψηφιστεί. Πάμε στο συμβιβασμό 10, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα τώρα. Υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα της 10, συμβαστικής 10. Υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίθηκε. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει, πολύ καλά. Περνάμε στην 114 και γυρίσαμε σελίδα. Όσοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 119 υπέρ, κατά, αποχές, συγγνώμη, μια στιγμή. Να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 114. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 114. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 114 ψηφίζουμε. Καταπίπτει λοιπόν. Πάμε στην 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 14 υπέρ. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές. Συμβαστική 14 εγκρίθηκε. 215 ως προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 218 και οι 222. Αποσύρθηκαν αυτές. Εντάξει, Συμβαστική 15 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές συμβαστική αυτή να το ελέγξουμε τώρα σε σχέση με το αποτέλεσμα συμβαστική 15 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά μάλιστα καταπίπτει η 15 πάμε στην τροπολογία 159 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 48 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 55 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Η 151 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Πάμε στην 223 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 224 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 225 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει και 226 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 20 υπέρ 18 εναντίον μία αποχή σας ευχαριστούμε. Um, Mrs. Κυρία Γκέπαρτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά και τον τρόπο με τον οποίο με τη δική μας ομάδα συνεργάστηκε. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες κόκκινες διαχωριστικές γραμμές που έχουμε εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα ιδιαίτερα όσον αφορά την τον πραγματικό συνολικά, την πραγματική εξαίρεση όσον αφορά τις υπηρεσίες και το θέμα του θετικού καταλόγου που δεν προχώρησε, δεν πέρασε και το θέμα για μια πρόταση που έγινε πώς το ESDS δηλαδή με άλλο τρόπο, με καλύτερο τρόπο θα πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε δεδομένες αρχές. Αυτά τα θέματα δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά και γι' αυτό για μας ήταν ανέφικτο, αδύνατο να εγκρίνουμε αυτή τη γνωμοδότηση ως ομάδα. Πράγμα το οποίο μας θλίβει ιδιαίτερα, γιατί θα θέλαμε να υπήρχε μια πολύ σαφέστερη τοποθέτηση από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή για αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα προστασίας καταναλωτών. Ευχαριστώ. Thank you very much. And, um, Ευχαριστούμε πολύ για την επεξήγηση αυτή. Και κάποια από τα σημεία που αναφέρατε αναγκαία σε σχέση με τις αρμοδιότητες της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής σίγουρα θα συνεχίσουν αυτά τα θέματα να μας απασχολούν σε σχέση με ε, τις αυθεντικές ε, αρμοδιότητες της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Κρίμα είναι ότι δεν μπόρεσε να υπάρξει μια συντριπτική πλειοψηφία. Είμαι βεβαία όμως ότι πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις θα διεξαχθούν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και να προχωρήσουμε καλύτερα. Και ευχαριστώ που μας επεξηγήσατε για τις διαχωριστικές γραμμές από την ομάδα σας που ήταν πολύ επικοδομητικό. So, Λοιπόν, επόμενη ψηφοφορία. Σελίδα 8 του καταλόγου ψηφοφορίας. Τροπολογία 131. του κυρίου Κριστιαν Σίλβιου Μπουσόη θα γίνει χωριστή ψηφοφορία. Δεν καλύπτεται από τη συμβαστική 13 η 131. Η Σίγητρα λοιπόν είπε ότι αυτή την τροπολογία 131 θα πρέπει να την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Δεν εντάσσεται στην συμβιβαστική. Το λέω αυτό ως διευκρίνηση πρωτού ξεκινήσουμε. Επίσης έχει αποσυρθεί από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Αλεξάνδρο, Αλεξάνδρο Μωράτη έχει αποσύρει την τροπολογία 42. Προσπαθώ να τη βρω. Είναι στο τέλος του καταλόγου. 42. Η Λάρα. Θέλω να πω το εξής. Όσον αφορά τον κατάλογο του ΕΛΚ, στο 116 υπάρχει κάποιο λάθος. Εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης Μπουζόη. Αυτό για το ΕΛΚ. Τώρα, αν θέλουν κάτι άλλο σοσιαλιστές, εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε σχέδιο γνωμοδότησης από την Λάρα σε σχέση με πρόταση οδηγίας για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτουν των εμπορικών απορρίτων κατά της παράνομης απόκτησης χρήσης και αποκάλυψής τους. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται. 25 προς 13. Τροπολογία 73. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένα έχει απορριφθεί. Έχει αποσυρθεί, συγγνώμη. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Σεβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μάλλον συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές Δεκτή. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε τροπολογία 2. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Την 86 παρακαλώ. εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε παρακαλώ. Τροπολογία 95. εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 98 υπέρ, 98 και 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε. Τροπολογία 106. Λυπάμαι, είχατε δίκιο, απορρίπτεται. Πρέπει να προσέχονται, μου λέει γραμματεία. Τροπολογία 107 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 108 υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 108. είναι σαφές ότι απορρίπτεται 109 α, καλύπτονται πάμε στην τροπολογία 3 υπέρ τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 111 όχι όχι καταπίπτει συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα τώρα πηγαίνουμε στην τροπολογία 131. Η τροπολογία που σας είπα πριν ότι δεν καλύπτεται και την ψηφίσουμε ως προσθήκη. Σας το είχα πει και από την αρχή, κάπου στην σελίδα 8. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ε, Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 149 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμπιβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, υπέρ 155, κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 15 που συνδέεται με την συμβαστική 4 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και 166 ε, που ήταν ταυτόσημη έχει γίνει δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 170 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 171 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 9 υπέρ, κατά να ελέγξουμε. Όχι, όχι. Η 9 εγκρίνεται. Η 9 εγκρίνεται. Πάμε στην 176 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά 177 πρέπει να την ελέγξουμε εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές όχι συγγνώμη καταπίπτει. Άρα που πάμε στην συμβαστική 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα 186-187 από κοινού τώρα είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 188 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 13 είναι γλωσσική φύσεω. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πρώτο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για τη διαγραφή του σημείου α υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, α, κατά πίπρι αν εγκριθεί προφορική τροπολογία. Πάμε στην 197 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 200, πίπτη. 201 έχουμε πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα όμως έχει αποσυρθεί. 203 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε τη 206 παρακαλώ. Απορρίπτεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 22 συμβιβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221. 221 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 222 και 223 υπέρ αυτών κατά αποχές καταπίπτουν. 224 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 225 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 226 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε. 226 παρακαλώ. That's fallen by one vote. Για μία ψήφο διαφορά πίπτη. 227 τώρα υπέρ κατά αποχές πίπτη. Εξετάζω να δω μήπως μπορούμε ομού να ψηφίσουμε πολλές τροπολογίες την 17 έως την 30. Από την 17 έως 30 μπορούμε να τις ψηφίσουμε ομού όλες. Όχι, όχι λέτε. Εντάξει λοιπόν. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι κάπου μπορούμε να προχωρήσουμε. Μία κάθε φορά. 17 λοιπόν τότε υπέρ κατά αποχές πίπτη. 18 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 19 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 20 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 23 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 24 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 21 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 22 υπέρ κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 22 και άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 26 τώρα υπέρ, κατά, αποχές. Καταπίπτει 25 υπέρ, κατά, αποχές. Καταπίπτει 27 υπέρ, κατά, αποχές. Καταπίπτει 28 υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει 29 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 30 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 35 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 3 συγγνώμη συγγνώμη 35. Να ελέγξουμε. Ξαναψηφίζουμε την 35 ηλεκτρονικά. 35. Ψηφίζουμε. 35 λοιπόν. Αυτή είναι που ψηφίζουμε. Μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε αυτή την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 35 και πάλι παρακαλώ. Εντάξει. Η τροπολογία 35 κατέπεσε. Τροπολογία 36 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. Πολύ καλά. Ελέγχουμε, ψηφίζουμε την 36. 36 λοιπόν. Εγκρίθηκε η 36. Ωραία. Η 37 υπέρ. Κατά. Από. Θα ελέγξουμε ξανά την τροπολογία 37 και αυτή θα την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. 37. Λοιπόν, κατέπεσε αυτή. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Τροπολογία 38 κατέπεσε. Η 40 κατέπεσε. Η 41 τώρα υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 42 αποσύρθηκε η 42. Η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 44 υπέρ κατά Συγγνώμη, εδώ λέει αν εγκριθεί κατέπεσε. Η 44 λοιπόν κατέπεσε. Συζητώ συγγνώμη. Δεν την ψηφίσουμε. Συμβαστική 4. Υπέρ. Α, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Πολύ καλό που μου το υπενθυμίσατε. Την καλύψαμε μέσω συμβιβασμού 15. Προχωράμε κατευθείαν στη 51 τροπολογία λοιπόν. Εντάξει, 51 τώρα τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 52, συγγνώμη. 53, σωστό, 53 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Ή 54 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. 55 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Ή 56 υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει. Η 57 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Η 58 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πέρασε και εγκρίθηκε αλλά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 58 ηλεκτρονικά άρχεται 58 λοιπόν η 58 κατέπεσε 59 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η 60 αποσύρθηκε 60 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 63 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 63 ελέγχουμε και ψηφίζουμε την 63 ηλεκτρονικά άρχεται και αυτή καταπίπτει με μία ψήφο διαφορά. 62 τώρα υπέρ κατά να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 62 ξανά ηλεκτρονικά. Σχεδόν τα καταφέραμε και τελειώνουμε. 62 λοιπόν άρχεται. Μία ψηφοφορία ακόμα έχουμε και ολοκληρώνουμε. Πέρας ψηφοφορίας 62. Καταπίπτει με δύο ψήφους διαφορά. 64 τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα ελέγξουμε και την 64 ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε. 64. 64. Αυτή ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Η 65 τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Καταπίπτει. 66 καλύφθηκε ήδη. Οπότε διεκπαιρεώθηκε, διευθετήθηκε. Περνάμε τώρα στο, στην ψήφιση της τελικής μορφής της έκθεσης ως έχει. Του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Παρακαλώ δύο ακόμα πρέπει να συμμετάσχουν. Ευχαριστώ. Και αποτέλεσμα Μάλιστα, εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια θερμά προς τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Κάποιες από αυτές τις ψηφοφορίες είχαν πολύ μικρή διαφορά ψήφων. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω μόνο ήθελα τους συναδέλφους και όλους τους εισηγητές και τα λοιπά. Ένα, ένα θαύμα σχεδόν καταφέραμε όσον αφορά τις προθεσμίες. Δεν έπρεπε να αναβληθεί τίποτα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία όλων.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 για θαύματα που έγιναν στον χρόνο σχετικά με την κυρία Ντυρόν. Η κυρία Ντυρόν είναι μία πρόταση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις. Η 36 παρακαλώ είναι η πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 37 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 37. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 37. Και άλλοι τρεις, παρακαλώ, πρέπει να ψηφίσουν Λοιπόν, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 6 σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 46, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 49 υπέρ κατά ε, μισό λεπτό ελέγχουμε ε, ηλεκτρονικά τη 49. Η τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 57 λάθος. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 60 υπέρ κατά αποχές ε, η 3 συμβαστική υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, η συμβαστική 4 εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 9, η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 11, όχι μισό λεπτό, έχει καταπέσει η 78 καταπίπτει, στην 80 πάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Η τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 83 νομίζω ότι εγκρίθηκε. Η 83. Εγκρίθηκε. Η 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 85 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι η 85 απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 85. Ελέγχουμε την 85. Η 85 εγκρίθηκε. Η 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. οι 87 υπέρ κατά εγκρίνεται. οι 88 υπέρ κατά εγκρίνεται. οι ε, 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 90 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 91 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 92 διαγραφή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 93 είναι διαγραφή και η 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 95 95 υπέρ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση 95. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας το 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται η 16 εγκρίνεται η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική η 2 και η 3 σε τμήματα πρώτο κομμάτι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα, μισό λεπτό. Όλα τα άλλα έχουν καταπέσει μέχρι τη συμβιβαστική 8. Λοιπόν, συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται, η 30 υπέρ κατά εγκρίνεται, η 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 32 παρακαλώ. 32. 32. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Η 33 απορρίφθηκε. Η 3 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι η 3 έχει εγκριθεί, αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχω με την τροπολογία 3. εγκρίθηκε η 34 υπέρ α, όχι έχει καταπέσει και τώρα ε, τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης ως τροποποιήθηκε Ευχαριστώ πολύ εγκρίθηκε 30 με 6 το αποτέλεσμα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 Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και θα προεδρεύσω εγώ μέχρι να επανέλθει πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Ζερι Ποσιπίση από το ΕΛΚ. Κύριε Πόπιζιλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω τον κανονισμό του Συμφουλίου και του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μειωδικά κινητά μηχανήματα πολύ τεχνικός ο τίτλος, ε, αλλά από νομικής πλευράς ουσιαστικά τα πράγματα είναι απλά. Περιδίνως πρόκειται για όρια εκπομπών ε, για τους ε, κινητήρες καύσης οι οποίοι τοποθετούνται σε εξοπλισμούς μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται στο δικό δίκτυο, στο δρόμο σε οδικά δηλαδή μηχανήματα. Στην πρόταση κανονισμού πρώτα απ' όλα ορίζεται ότι ε, διέπεται από αυτά τα μη οδικά μηχανήματα. Πρόκειται για πολλά είδη εξοπλισμού, φορητά μηχανήματα, μικρά, μέχρι και σιδηροδρομικούς σειρμούς ε, και άλλα πιο πολύπλοκα μηχανήματα δεν είναι κάτι καινούριο. Ουσιαστικά είχαμε και την οδηγία 98 κάθετος 68 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτή συνδέεται αυτό ο κανονισμός. Αυτή η οδηγία έχει τροποποιηθεί αρκετέ φορέ κατά το παρελθόν. Γενικά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ενδεδειγμένη, διότι δεν κάλυπτε ένα μεγάλο αριθμό κινητών μηχανημάτων και διάφορα είδη κινητήρων. Εξού και αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια νέα πρόταση που πρέπει ουσιαστικά να νομοθετήσει καλύτερα τα όρια εκπομπών αυτών των κινητήρων που δεν καλύπτονταν πριν. Έχετε λοιπόν τους ορισμούς, τους νομικούς ορισμούς στην αρχή και αν δείτε τις τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει ως εισηγητής, θα διαπιστώσετε ότι διευρύνω τους ορισμούς αυτούς. Παραδείγματος χάρη, περιλαμβάνω τους κινητήρες αντικατάστασης. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα. Έχω λάβει μέρος προσωπικά σε πολλές συζητήσεις που αφορούν ακριβώς το θέμα αυτό. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό ο κανονισμός μεταξύ, ε, μάλλον ε, εντός αγωγικών θα μπορούσε να βλάψει κατασκευαστές ε, ή φορείς οι οποίοι συνεργεία που αντικαθιστούν κάποιους κινητήρες. Και γι' αυτό και κατέθεσα την τροπολογία για τον κινητήρα αντικατάστασης, ας πούμε, σε κάποιες ατμομηχανές, σε κάποιους συνδεδραμικές μηχανές. Πολλές φορές πρέπει να αλλάξει ο κινητήρας. Το στις συνδρομικές στις μηχανές υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αλλάξει ο κινητήρας. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι αν έχουμε ένα ήδη υφιστάμενο μηχάνημα και απλά καθιστούμε τον κινητήρα, δεν θα πρέπει ο κανονισμός να καλύπτει αυτού του είδους την περίπτωση. Άλλες είναι οι παράμετροι των νέων κινητήρων. Και βέβαια είναι δύσκολο. να τοποθετηθούν σε υφιστάμενα μηχανήματα οι νέοι κινητήρε. Γι' αυτό μιλάμε για κινητήρε αντικατάσταση. Ζητούμε δε παρέκκληση. Όλε οι τροπολογίε έχουν ω στόχο την προστασία του περιβάλλοντο αφενό, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αφετέρου, αλλά και να έχουμε έναν κανονισμό που να μπορεί να εφαρμόζεται στην πράξη. Έτσι οι κατασκευαστές θα μπορούν, θα έχουν το χρόνο στη θέση τους για να καταρτήσουν τις παραμέτρους του νέου προϊόντος. Αν τεθεί σε εφαρμογή πάρα πολύ γρήγορα αυτή η νομοθετική πρόταση θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητες αντιδράσεις των κατασκευαστών. Αυτό είναι ένα θέμα. Και άλλο ένα θέμα είναι η Χρήστε ή οι φορείς εκμετάλλευσης. Σας είπα το παράδειγμα ενός σειρμού με τη σιδηροδρομική μηχανή. Εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί ε, ο κινητήρα αυτή τη δρομική μηχανή, θα πρέπει να μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτό, που είναι πολύ δαπανηρό, φορεί εκμετάλλευση, με τον κινητήρα αντικατάστασης όπως τον λέμε, και όχι να χρειαστεί να αλλάξουν όλη τη μηχανή τη συνδεδρομική και να αγοράσουν μια καινούργια. Άρα προστασία περιβάλλοντος, συμφέροντα χρηστών, συμφέροντα των κατασκευαστών. Μιλάμε άλλωστε για πολύ δαπανηρό εξοπλισμό. Σας ανέφερα πλιστάκι στο παράδειγμα των συνδρομικών μηχανών και οι κατασκευαστές τέτοιων μηχανών μου είπαν ότι πολλές φορές στη διάρκεια του κύκλου ζωής ε, μια μηχανή χρειάζεται να αντικατασταθεί ο κινητήρα. Και φυσικά οι φορεί εκμετάλλευση πάρα πολύ δύσκολα μπορούν ε, να αλλάξουν όλο το σειρμό, ε, όλη την ε, μηχανή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δαπανηρό αυτό. Άρα δεν είναι και τόσο δύσκολο και πολύπλοκο από νομικής πλευράς. Το θέμα, εγώ στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια ξεκάθαρη βούληση από πλευρά τη να προτείνει μια καλύτερη νομοθετική πρόταση και για τις εκπομπές της αερίων. Γιατί αυτή η πρόταση δεν αφορά μόνο τον όγκο, και την ποσότητα των σωματιδίων, αλλά και τη μάζα των σωματιδίων. Λαμβάνουμε δηλαδή καλύτερα υπόψη την επικινδυνότητα των ρήπων για το περιβάλλον. Άρα η οδηγία βελτιώνεται με αυτή την νομοθετική πρόταση. Αυτά λοιπόν είναι δισαγωγής. Η πρόταση αυτή πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση, γιατί στόχος είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και η καλύτερη ρύθμιση, ιδίω για όσους ε, θα κάνουν χρήση αυτού του κανονισμού. Υπάρχει επίσης η βούληση να μην θυγούν, ε, να μην πηγούν οι φορείς εκμετάλλευση τέτοιων εξοπλισμών και να εξευρεθεί μια συμβαστική λύση με τους κατασκευαστές. Αυτά και προσβλέπω να έχω μια καλή συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ στον, τον εισηγητή. Πολύ συνοπτικά και με πλήρη τρόπο μας παρουσίασε τα πράγματα. Έχουμε διάφορους σκιώδεις εισηγητές. Η Μαρία Γκραπίνη είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο από την ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θερμά συγχαρητήρια προς τον εισήγητη. Δυσχερές το θέμα της έκθεσης και τεχνικού χαρακτήρα. Όμως ταυτόχρονα έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι ίδια μηχανολόγος και έπρεπε να διαβάσω αρκετά κείμενα για να κατανοήσω προς τα που θα μας οδηγούσε η αναθεώρηση της οδηγίας, η αναδιατύπωση αυτή τις προτάσεις του εισηγητή και τις δικές μου τροπολογίες τις ανέλησα. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν πρόσθετα κόστη, πρόσθετες δαπάνες. Στους κινητήρες αντικατάστασης είναι καλή πρωτοβουλία κινητήρες αντικατάστασης ή αμοιβή κινητήρες να χρησιμοποιούνται ώστε να μην αλλάζει ολόκληρο το όχημα όπως ε, μια οτομοτρής για παράδειγμα, ένα τρένο. Έχουμε ένα πρόβλημα όμως, πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση, να δούμε πώς μπορεί να πετύχει μια τέτοια αντικατάσταση κινητήρα να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή κινητήρες που από το 2011 θα έχουν παραχθεί. Πώς μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια θα διασφαλίζεται για τον χρήστη αφενός και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ρήπανση του περιβάλλοντος θα είναι μειωμένη. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε μεταχειρισμένους αμοιβού κινητήρες αντικατάστασης όπου θα ρηπαίνουν το περιβάλλον και θα ρηπαίνουν περισσότερο κιόλας από ότι ο αρχικός κινητήρας ο οποίος αντικαθίσταται. Ο εισηγητής προτείνει το άρθρο αυτό να διαγραφεί. Πρόκειται για το θέμα της συμβατότητας εδώ, να δούμε αν συνάδει αυτό ή όχι. Και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις που θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Η απόλυτη διαγραφή του πιστοποιητικού συμβατότητας δεν νομίζω ότι είναι σωστό, σωστή υπόθεση διότι μέσω ενός τέτοιου πιστοποιητικού μπορεί κανείς ε, να ενισχύσει την λειτουργία αυτών των ε, κινητήρων. Να μην διαγραφεί λοιπόν, αλλά να αναδιατυπωθεί αυτό το εδάφιο. Τελευταία σκέψη. Και το άρθρο 46, να μην ε, διαγραφεί πλήρως. Υπάρχουν εσωτερικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν αυτού του είδους την λειτουργία. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την διασφάλιση της πτυχής προστασίας καταναλωτών. Πρόκειται για δοκιμές, δοκιμές λειτουργίας κινητήρων. Δεν πρέπει να διαγραφεί, πρέπει να διασφαλιστεί, να διατηρηθεί. Θα καταθέσω τροπολογίες για αυτό το θέμα και ελπίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια έκθεση στην οποία θα καταλήξουμε, η οποία θα βελτιώνει το υφιστάμενο πλαίσιο και το, τα όσα ισχύουν για αυτές τις ε, κινητές συσκευές ε, και κινητήρες. Ευχαριστώ. Και τώρα έχετε εσείς τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα υποστηρίζουμε τη γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πλουστευτεί η νομοθεσία, να είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί και να υπάρχει βελτίωση και του ατμοσφαιρικού αέρα. Είχα κάπως ένα ερωτηματικό τι γίνεται σε σχέση με τέτοιου είδους αντικαταστάσεις Πολλές φορές πρέπει να υπάρχουν πολλά δικαιολογητικά. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ή όχι. Θέλω να πιστώ λίγο παρα, παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, η ευθυγράμμιση των ορίων όσον αφορά τους ρήπους για την ΕΕ και τη ΣΥΠΑ είναι σημαντική υπόθεση και πρέπει να ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις που έχουμε με τη ΣΥΠΑ για την TTIP, τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου. Για κάποια από τα συγκεκριμένα θέματα για τους ρήπους όσον αφορά πλωτές οδούς για παράδειγμα, ιδιαίτερα για υψηλότερης υποδύναμης κινητήρες, Υπάρχουν εδώ φόβοι ότι ίσως θα υπήρχαν κάποιες απρόβλεπτες επιπτώσεις που δεν θα θέλαμε να ε, επισυμβούν. Δεν θέλουμε να έχουμε υπερβολικούς τρύπους. Θέλουμε να έχουμε ισόρροπη προσέγγιση, να βελτιωθεί ο ατμοσφαιρικός αέρας. Από την άλλη πλευρά να μην εξωθηθούν εκτός ευρωπαϊκής αγοράς κάποιες επιχειρήσεις. Καλωσορίζω λοιπόν τις τροπολογίες για την αντικατάσταση κινητήρων ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται αυτή η λειτουργία ε, κινητήρων αντικατάστασης όπως και στα ΙΟΤΑΣΥ για παράδειγμα όταν έχουμε και δυσανάλογο για παράδειγμα ποσοστό κινητήρων diesel εσωτερικής καύσης είναι λοιπόν σωστό οι μικροί, ε, μικρής εμβέλειας ε, χρήστες να ληφθούν υπόψη και σε σχέση με μια βλάβη μηχανής να μπορούν να βοηθηθούν να αντικαταστήσουν το υψηλό κόστος που συνεπάει την αντικατάσταση ενός ολόκληρου μηχανισμού ή με αντικατάσταση κινητήρων και η μεταβατική περίοδος να ισχύει για έξι μήνες ώστε να έχουν το χρονικό διάστημα οι εταιρείε να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ για, τους, ε, για την προσπάθεια του εισηγητή και των σκιωδών. Sorry, didn't have the microphone I want to Ήθελα να δώσω το λόγο και στους φιλελεύθερους, αλλά δεν είναι παρόν ο σκιώδης συγητής. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο σκιώδη συγητή από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό νομίζω ότι ίσως μπορώ να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποια προκαταρκτικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων μεταξύ ε, εισηγητού και επιτροπής και σε ό,τι αφορά τους στόχους για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους για τη λειτουργία της εσωτερική αγοράς και κυρίως όμως για τους στόχους ε, σε ό,τι αφορά την απλούστευση και την αποτελεσματικότητα των, ε, της νομοθεσίας. Και πάνω σε αυτά θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Όλοι αναγνωρίζουν ότι ένα το σημείο της φυστάμενης οδηγίας ήταν η δυσκολία εφαρμογής, αποτελεσματικής εφαρμογής. Ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, που διατίθενται στο εμπόριο, συμμορφώνονται πλήρως με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα όρια εκπομπών, για την ε, ποιότητα του αέρα. και ασχοληθήκαμε με το θέμα και προτιμήσαμε να υποβάλουμε πρόταση κανονισμού ώστε οι κανόνες να είναι συγκεκριμένοι και να ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλείο όπως αυτό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για να μπορούμε να επαληθεύουμε ότι έχουμε τα στοιχεία που ε, μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι μόνο συμβατά με όλους αυτούς τους κανόνες μηχανήματα κυκλοφορούν ε, στο εμπόριο. Είχαμε κάποιες συζητήσεις και με την Επιτροπή σας γιατί εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε τα εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή αλλά να έχουμε μια συζήτηση για την πρακτική εφαρμογή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Αυτό ως προκαταρκτικό σχόλιο. Ευχαριστώ. Μήπως ε, θέλετε κάτι να πείτε κύριε Σιγητά για να απαντήσετε στους εσκιώδεις ε, και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Πράγματι υπάρχει σύγκληση απόψεων, είναι κοινή φιλοσόφια που δέχεται δύο προτάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας να διευκρινίσουμε τον ορισμό για τον κινητήρα αντικατάστασης. Θα επαληθέσω αυτά που είπατε. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 46, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Ε, ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή βέβαια. Εγώ είμαι ανοιχτό όμως να το συζητήσουμε. Και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα όρια, προσπάθησα να έλθω σε επαφή με τους κατασκευαστές ε, των διαφόρων ειδών εξοπλισμού, <clears throat> μικρών φορητών μηχανημάτων ή μέχρι και τους κατασκευαστές ελκυστήρων και ε, σειροδρομικών μηχανών. Και όλοι συμφωνούν ε, με τη σκοπιμότητα της μείωσης αυτής των εκπομπών. Το ερώτημα που είναι μήπως όμως οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές θυγούν με αυτόν τον κανονισμό. Εγώ δεν διαπιστώνω κάτι τέτοιο. Τα όρια εκπομπών δεν θεωρούν οι κατασκευαστέ ότι αυτό μπορεί να αποβεί σε βάρος τους. Θα τα σεβαστούν αυτά τα όρια. Το πρόβλημα είναι το χρονοδιάγραμμα η περίοδο εφαρμογή. Ε, γιατί τότε πρέπει να προε... για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να προετοιμαστούν οι κατασκευαστές ώστε τα προϊόντα που θα διαθέσουν στο εμπόριο να ε, συμμορφώνονται με του νέου κανόνε. Αυτά προ το παρόν. Να συζητήσουμε λοιπόν τι τροπολογίε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you, ε, Rapporteur. Just to go over the deadline for amendment. Ας δούμε λοιπόν τι καταληκτικέ ημερομηνίε για τροπολογίε 14 Απριλίου. Η τροπολογίες ε, ε, θα πρέπει να εξεταστούν 6-7 Μαΐου και 22 Ιουνίου η ψηφοφορία ε, στις 23 Ιουνίου. Προφανώς πρόκειται για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστούμε τους Σκιώδης, τον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επόμενο τώρα θέμα της ημερήσιας διάταξης Η κυρία Γκέπχαρτ ε, ίσως ε, μπορεί ε, να αναλάβει την Προεδρία για να παρουσιάσω και εγώ τη δική μου έκθεση. Νομίζω ότι είναι το παλαιότερο μέλος σε αυτήν την Επιτροπή. Okay. Χωρίς να έχω προετοιμαστεί το κάνω αυτό και συγγνώμη αν κάπως ε, κάποια πράγματα δεν πάνε με τον ε, αναγκαίο ρυθμό. Περνάμε τώρα σε σχέση με τις συσκευές ε, αερίου, καύσης αερίου. Η συγκίτρια η κυρία Στάιλερ. Έχει τον λόγο, Κάθριν, παρακαλώ. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ, Πρόεδρε. To, uh, Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Όπως εισήγαγα το θέμα της έκθεσης κάποιες εβδομάδες πριν, είναι μεγάλη σπουδαιότητα στο χαρτοφυλάκι όσον αφορά την ασφάλεια. Επίσης και όσον αφορά και πρέπει να το θυμόμαστε ότι 40 δις είναι ο τζίρος για την χρήση αυτών των συσκευών 1,7 για, τις, ε, για την, ε, τα κάψιμα και 40 δις ε, για τις συσκευές. Έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για την ασφάλεια το θέμα αυτών των μηχανών συσκευών και με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, 27 τροπολογίες από τους συναδέλφους, να τις πάρουμε αυτές τις 27 τροπολογίες, να τις δούμε. Κάποιοι είναι παρόντες από τους συναδέφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες στην 202, 203, 204 τροπολογίες. Είμαι βεβαίω ότι μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό για αυτές. Για την τροπολογία 205 επίσης, και εκεί βαίνει καλός θα λέγα, είναι εδώ και η δική σου τροπολογία, Ντίτερ, που είναι και αυτή σημαντική για την 216, 209, Βαίνουν, βαίνει καλός. Αν πάμε στην 210, δείτε μια από τις δικές σου, το τελευταίο τμήμα της πρότασης που λέει ε, εξαιρέσεις, ε, ίσως θα πρέπει να αποσαφινιστεί κάπως αυτό. Τι συμβαίνει δηλαδή σε σχέση με το εύρος και την λειτουργία όσων θα ενταχθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το σημείο εξειδικευμένα. Αν πάμε τώρα στην 211 τροπολογία, προφανώς εδώ πρόκειται για ένα νέο ορισμό που θα χρειαζόταν. Πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει νομική σαφήνεια για την 211, την 212, 213 και 214 ίσως επίσης και για αυτές. Όλες αυτές μπορούν να συνεξεταστούν λοιπόν και αν δούμε τη 215 που είναι το αντικείμενο αποσαφηνήσεων που χρειάζονται, θα μπορούσα να εξετάσω το αίτημα. Για την 216 βαίνει καλός, η 217, η 218 μέχρι και την, τις τροπολογίες στη συνέχεια μια στιγμή να το κοιτάξω ξανά Λοιπόν, από τη 16 έως τη 226 νομίζω βαίνουν καλώς και μπορώ να τις δεχτώ. Για 227 χρειάζομαι αποσαφήνιση, χρειάζομαι διευκρινήσεις. Και την 228 εντάξει πάλι, αλλά η 229 θέλω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ τους συναδέφους που ανάλωσαν χρόνο για να προσθέσουν κάποια στοιχεία στα όσα είχαμε εμεί εκπονήσει. Πρόκειται για μια πρόταση που ευθυγραμμίζει τα όσα θα, θα λειτουργήσουν. Αυτό που θέλουμε είναι να ενισχυθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν τα πράγματα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προσπάθεια να προσθεθούν αυτά τα στοιχεία και πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις των προστιθέμενων τροπολογιών εδώ. Είμαι βεβαίω ότι μπορούμε να εξεύρουμε τροπολογίες συμβιβαστικέ, οπότε λοιπόν ε, εκείνες που δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή πλήρως αυτή τη στιγμή ζητώ νομική αποσαφήνιση για το τι συμβαίνει. Ζητώ λοιπόν να αποσαφινιστούν κάποια σημεία ελπίζοντα ότι θα μπορεί να βρεθεί λύση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Μπουσόη, σκιώδη από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και με την άδειά σας μια και πρόκειται για τεχνικό θέμα σε αυτή την έκθεση, θα μιλήσω ρουμανικά για να είμαι βέβαιος ότι θα συνεννοηθούμε σωστά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κυρία Στάιλερ για τις παρατηρήσεις σας. Σίγουρα. Ήδη το προαναφέρατε αυτό και έχω καταθέσει τροπολογίες κι εγώ και θα ήθελα επ' αυτό να τονίσω τα εξή στοιχεία. Πολύ σύντομα βέβαια. Στην 204 για τον κανονισμό. Ο κανονισμός δεν πρέπει μόνο να αναφέρει ένα κάποιο κίνδυνο του μονοξυδίου του άνθρακα, αλλά θα πρέπει να εξετάζει και την ασφάλεια των καταναλωτών, ώστε μια συσκευή να ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες. Υπάρχουν και άλλες βλαβερές εκπομπές ρήπων και άλλες, ε, άλλοι ρήποι οι οποίοι έχουν αρνητική επίπτωση στους, ε, στην υγεία των καταναλωτών. 206. Να υπάρξει ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους πολίτες όσον αφορά την ανάγκη συντήρησης αυτών των συσκευών ώστε να αποφευθούν πιθανοί κίνδυνοι ή οποιασδήποτε βλάβες και προβλήματα. Άλλες τροπολογίες από κοινού με την κυρία Μπουνόβα έχω καταθέσει. Θα έλεγα και ο εξοπλισμός ε, θα πρέπει να προβλέπει μια, ας ένα ενιαίο πιστοποιητικό λειτουργίας ή συμβατότητα. Στη δική μου χώρα, τη Βουλγαρία, είναι δύσκολη υπόθεση να υποβάλλονται διαφορετικά τέτοια πιστοποιητικά συμβατότητας. Λοιπόν, το θέμα του πιστοποιητικού συμβατότητας αν είναι ενιαίο, θα εξαπλουστεύσει πολύ, θα απλουστεύσει τον τρόπο λειτουργίας και θα μπορεί να επαρκεί πλήρως 211 και 212. Εδώ κάποιους ορισμούς εισάγω με τις αναγκαίες λεπτομέρειες και εξειδικεύσεις για την ποιότητα των αερίων με την οποία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σωστά και φιλοπεριβαλλοντικά ένας κινητήρας. Την 213 την απέσυρα, 226 τώρα. Και όσον αφορά ε, για παράδειγμα εδώ μια ψυχολογική, ένα ψυχολογικό στοιχείο για τις, ε, για, για τις ε, τη συμπίεση αερίων από πλευράς δοχείων συμπίεσης και για την 229 έγκριση τύπων όσον αφορά την τυπολογία συσκευών. Τα έχουμε λάβει υπόψη αυτά ώστε να μπορέσουν όλα να λειτουργήσουν σε ένα σωστό πλαίσιο. Αν θα έχει συγκεκριμένη διορία ένα τέτοιο πιστοποιητικό θα περιτεύει αυτό. Μία είναι η πτυχή της πιστοποίησης Άλλο όμως είναι η επιτήρηση και εποπτεία των συσκευών αυτών που θα διοχετεύονται στην αγορά και γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτό να το δούμε και ξεχωριστά. Thank you. Dan Dalton for the ECR. Thank you, Chair. Dan Dalton από την ECR. Ε, κοιτάξτε, προφανώς όλα αυτά πρέπει να είναι λειτουργικά. Και επειδή πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό χαρτοφυλάκιο, δεν έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες και αυτό δείχνει ότι υπάρχει συμφωνία για το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Εγώ έχω δύο θέματα που θέλω να δείξω. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να προφέρουμε ένα σύστημα για να μην υπάρχει υπερβολική βαθμολογία. Δεν νομίζω ότι θέλουμε ε, μία που να ταιριάζει βέβαια παντού, άρα δηλαδή θα πρέπει να εξετάσουμε ε, την ε, καινούργια βαθμολογία οπουδήποτε είναι κατάλληλη και δεν μας απομακρύνει από την νομοθεσία. Και να πω και αυτό που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής ότι οι τροπολογίες για το μονοξίδιο του άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το ελέγχουμε. Όμως δεν είναι το μόνο θέμα ασφαλείας ε, που έχει σχέση με αυτές τις συσκευές. Ε, δεν πρέπει να δώσουμε υπερβολική σημασία στο μονοξίδιο του άνθρακα και να αγνοήσουμε άλλους κινδύνους. Να υπάρχει μια ισορροπία. Κατά τα άλλα είμαι απόλυτα ευτυχής. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του, την εισηγήτρια μάλλον. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Βέβαια ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως ξέρετε εγώ έχω καταθέσει αρκετές ε, τροπολογίες, ε, θα εστιάσω σε τρεις εξ αυτών. Η πρώτη αφορά το μονοξίδιο του άνθρακα Νομίζω ότι όσον αφορά το κείμενο προσπάθησα να βρω ε, συμβαστική διατύπωση για την τροπολογία σας. Ε, νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα στο νομικό κείμενο ε, και μπορεί να είναι αποδεκτή αυτή η τροπολογία. Κατόπιν, αν πάμε στις βαθμολογίες πρέπει να συμπεριλάβουμε την διατύπωση αυτή που αφορά τις συσκευασίε και όχι τα ίδια τα προϊόντα. Αυτές είναι πραγματικά τεχνικές ε, τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικές. Και τέλος, όπως είπα και στην τελευταία συζήτηση, δεν ε, στηρίζω την απέτηση να υπάρχει ε, μόνο επαγγελματική συντήρηση. νομίζω ότι αρκεί μια σύσταση, αυτό μπορεί να είναι ένα είδους συμβιβασμού. Πασκάλ Τυρά από του ε, Πρασίνου δεν είναι παρόν. Δεν υπάρχει ούτε σκιώδη από την ομάδα FTD. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Θέλετε να ακούσουμε την Κομισιόν. Να ακούσουμε την Κομισιόν, παρακαλώ. Thank you. <clears throat> So, thank you for the report and for the... Ευχαριστώ και για την έκθεση και για τι τροπολογίε. Εμεί θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σα στην τροπολογία 211 στην τροπολογία 212, διότι εδώ οι ορισμοί δεν ανταποκρίνονται ε, στη δική μας αντίληψη. Ουσιαστικά αυτή τη διακύμαση ποιότητα του αερίου τη λαμβάνει υπόψη ο σχεδιαστής ε, της συσκευής αερίου και κοινοποιείται από την Κομισιόν. Δεν γίνεται ανάποδα αυτό, αντίστροφα. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί γίνεται αναφορά στη συμμόρφωση χωρίς νομικές πράξεις για τον ορισμό αυτό. Η τροπολογία 213 από ό,τι καταλάβαμε έχει αποσυρθεί, αλλά πάλι στη 212 η κανονική διακύμαση της ε, πίεσης και η ποιότητα του ε, κοινοποιείται από τα κράτη-μέλη και βάσει της προσαρμογής που θα πρέπει να υπάρξει για να είναι ασφαλή αυτά τα μηχανήματα, αυτές οι συσκευές. Θα πρέπει δηλαδή ο κατασκευαστής να προσαρμοστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τροπολόγες 210, 218 και 225 θα να σε, στη σήμανση αυτών των εξαρτημάτων. Η εξαίρεση ε, για τη σήμανση με το C ή είναι όταν δεν μπορεί να μπει στο εξάρτημα. Συμφωνούμε με την ατολική σκέψη, αλλά εμείς θα θέλαμε να προτείνουμε όταν μπουν αυτά τα σήματα. Στο άρθρο 18 ε, προβλέπουμε, έχουμε τους κανόνες για αυτή τη σήμανση C E. Και έχουμε την παράγραφο 1 για τις συσκευές, τη δεύτερη για την ε, τοποθέτηση του σήματος και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν να μπει στο εξάρτημα, τότε να μπαίνει στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής. Σε ό,τι αφορά τα 10 έτη για την τροπολογία 229. Εμεί προτείνουμε να παραμείνει η προθεσμία αυτή, γιατί έχουμε το θέμα της ανανέωση των πιστοποιητικών. Και υπάρχει και η 204 που δεν είναι ξεκάθαρη. Κάτι λέει για την ε, διαρροή των ε, συμπυκνωμάτων. Η ΣΥΓΙΤΑ θέλει να επανέλθει ναι, Ευχαριστώ. Είναι πράγματα αυτά ζητήματα που έχουμε να κάνουν με την ασφάλεια δικαίου. Ίσως μπορούμε να βρούμε συμφωνία για κάποια θέματα. Σε άλλα είναι μάλλον πιο προβληματικά. Το θέμα είναι να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά αυτά τα τεχνικά σημεία. Μια τεχνική πρόταση άλλωστε έχουμε ενώπιον μας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συναντηθούμε με τους σκιώδεις και να προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβεβαστικέ προτάσεις. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, υπάρχουν και οι αρμοδίδες των κρατών μελών, αλλά νομίζω ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή για να προχωρήσει αυτή η σήμανση, αυτή η πρόταση γιατί είναι σημαντική. Σημαντικό αυτό το νομοθέτημα για τις ε, συσκευές αερίου που επηρεάζουν τόσους πολλούς ανθρώπους, την ασφαλειά τους. Είναι η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων φυσικά ζωτική σημασία. Γιατί εκπροσωπούν και του καταναλωτέ στην Επιτροπή μα. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συνεργαστώ με του ε, σκιώδει. Δεν θέλω αν θέλετε να μας, ε, να υπενθυμίσετε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί εγώ δεν έχω μπροστά μου τις ημερομηνίε. Πρόεδρος, ναι, βεβαίω εξέταση συμβαστικών τροπολογιών 20 Απριλίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 23 Απριλίου, ελπίζοντας να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις το Μάιο και να ξεκινήσουμε έπειλα των Προεδρίας μάλιστα αυτές τις διαπραγματεύσεις σε ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει και άλλα θέματα. Θα δώσω ξανά το, την Προεδρία στην κυρία Στάιλερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση της Προέδρου μας, Βίκη Φόρτ, για τα μέσα ατομικής προστασίας. Η έχει το λόγο. Ευχαριστώ τους χειώδεις εισηγητές για την πολύ επικοδομητική συνεισφορά τους με τις προτάσεις τους. Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση στο Στρασβούργο και σε σχέση με τους άλλους σκιώδεις που δεν παρίστανται και πρέπει αν χρειαστεί να μπορέσουν και εκείνοι να ενημερωθούν. Υπάρχει συνένεση επί αρκετών θεμάτων και υπάρχουν κάποιες διστάμενες απόψεις. Συντάσσω συμβαστικές τροπολογίες σε τρεις κατηγορίες που θα έχουν ολοκληρωθεί κατά τα τέλη αυτής της ε, τρέχουσας εβδομάδας. Η μία κατηγορία αφορά το εύρος, ε, τα εδάφια 9 και 31 και το άρθρο 2, εδάφιο 2 τροπολογία 147 έως τροπολογία 151, 164, 167 και 180 έως την 255. Οι επόμενοι συμβιβασμοί θα είναι για την περίοδο ισχύω ε, και για την διαδικασία επικαιροποίηση. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις που κατέθεσε προτού εξεταστεί αυτός ο γύρος και κατηγορία τροπολογιών. Αυτός ο τομέας συμβαστικών τροπολογιών θα καλύπτει το, την αιτιολογική σκέψη 24, άρθρο 8, και θα είναι οι τροπολογίες 157 έως 160, 183, 184, 206 και 234 έως 238. Σε αυτόν τον τομέα συμβαστικών τροπολογιών η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ασφάλειας εξέθεσε σε μένα και τους κοιόδης ενδιαφέρουσες προτάσεις για μια πλουστευμένη διαδικασία και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών για τις προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφάλειας. Και καθώς οι συμβιβασμοί στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι τα θέματα θα, έχουν, θα εντάσσονται στη σωστή κατηγορία κινδύνων, <clears throat> παράρτημα 1, το 3 και τις τροπολογίες 217 έως 222, Έχουμε και έναν αριθμό κάποιων άλλων τροπολογιών που θα μπορούσα να υποστηρίξω, ιδιαίτερα όσον αφορά λεπτομέρειες λειτουργίας που θα πρέπει να βρίσκονται στη γλώσσα των κρατών μελών και όπου αποτελούν αντικείμενο εμπορία αυτές τις συσκευές 186, 188, 196, 230 και 231 τροπολογίες. Επίσης υπάρχουν προτάσεις ώστε να είναι τα σύμβολα ε, με τέτοιο τρόπο εφικτά και ηλεκτρονικά 193, 207, 227 και συναφείς τροπολογίες. Ένα εύρος πολύ επικοδομητικών τροπολογιών που αφορούν τις, ε, ε, τα επικολου, τις ετικέτες που θα πρέπει ε, να, ε, να δούμε ότι δεν αφορούν μόνο αποκλειστικά θέματα ασφάλειας. Τροπολογία 148, 175, 176, 177, Αρμό, Ροσφόρ και Μαστάλκα και να δούμε πώς θα μπορούσαμε ίσως να συνεργαστούμε για να ενταχθούν μέσα σε συμβαστικές τροπολογίες αυτές οι προτάσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες προτάσεις που μου δημιουργούν κάποιες ανησυχίες. Η 190 του κυρίου Μαστάλκα για ε, διάφορες ε, οδηγίες όπου αρκετοί εμπλεκόμενοι μου είπαν ότι θα δημιουργεί το μεγάλη σύγχυση για τους ενδιαφερόμενους. Αντί να υπάρξει απλούστευση θα ε, δημιουργεί το σύγχυση και με ανησυχεί αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην υπονομεύσουμε το έργο των συναδέρφων μας όσον αφορά την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα στις αγορές ε, αυτών των ε, ε, στοιχείων. Να δούμε τι γίνεται με την 192 και την 197. Ίσως είναι γλωσσικό ζήτημα και που ίσως θα μπορούσε να καλύπτεται από πλευράς τροπολογιών στη δέσμη που έχει κατατεθεί θα έπρεπε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τη διατύπωση όσον αφορά αυτό το πλαίσιο τροπολογιών. Θα ήθελα επίσης να μου, να μου πείτε πώς τα όσα η κυρία Άντερσον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε για το θέμα αυτό όσον αφορά την εισαγωγή της αρχής ε, της προφύλαξης, της αρχής της πρόνοιας διότι είπε λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι αναγκαία η αρχή της πρόνοιας και πρόληψης αλλά εδώ πρόκειται για εναρμόνιση και εδώ θα πρέπει πραγματικά να έχουμε πραγματογνωμοσύνη που θα μας καθοδηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες κατευθύνσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά προτάσεις, για παράδειγμα όπως την 166 για αυτή την έκθεση. Τροπολογία Ροσφόρ 210, 211, 212 που το καθιστά επιτακτική ανάγκη για τις, ε, τους φορείς ε, πιστοποίησης και αξιολόγησης να μπορούν να λειτουργούν μέσα σε πλαίσια εθνικής ε, συμβατότητας και πιστοποίησης. Υπάρχει εδώ το θέμα του ότι μπορεί να υπάρξει πρόσθετη αξία και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης από πλευράς κυρίου Πρέτσο έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες πράγμα το οποίο δεν θα σήμαινε ότι μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή έδρα ή όνομα θα έπρεπε να αναφέρεται από πλευράς παραγωγού θα μπορούσε να υπάρχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έρθει σε επαφή υπό αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση Ξέρω ότι αυτό αποτελεί λοιπόν μια παρέκκληση και ίσως θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ή όχι μπορεί να γίνει χρήση μιας τέτοιας ε, πρότασης. Τώρα, <clears throat> για την επόμενη συνάντηση σκιωδών θα είναι η 14η Απριλίου όπου θα ξανασυναντηθούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Η Σκιώδης. Ο πρώτος από πλευράς του ΕΛΚ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία εισηγήτρια, σας ευχαριστώ για όσα μας εκθέσατε σε, αυτή την, αυτό το γύρο, ας τον αποκαλέσω έτσι. Προσπαθούμε με αυτή την πρόταση δύο πράγματα να επιτύχουμε και το ένα από αυτά είναι στους καταναλωτές να προσφέρουμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τα όσα χρησιμοποιούν και να αποφύγουμε υπερρύθμιση, υπερβολικό επίπεδο ρυθμίσεων και διατάξεων ώστε επιχειρήσεις που δρούν σε αυτή την αγορά να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετες δαπάνες ή κόστη. Τώρα αναμένω και προσδοκώ, προσβλέπω τις συμβαστικές τροπολογίες που θα κατατεθούν. Σε σχέση με το Στρασβούργο τα πράγματα προς σωστή κατεύθυνση, με σωστό τρόπο τα συζητήσαμε και νομίζω ότι επί πολλών μπορεί να υπάρξει συμφωνία και να προχωρήσουμε. Για μένα και την δική μου πολιτική ομάδα είναι σημαντικό βέβαια εμείς σε δύο τομείς να μπορέσουμε να βρούμε θετικές συμφωνίες, συνενέσεις. Το ένα είναι το εύρος, το πεδίο εφαρμογής και ισχύω. Πρέπει επ' αυτού να βρούμε λογικούς ορισμούς τι θα είναι πέσα και τι όχι ώστε να υπάρξει μια νομική βεβαιότητα και ασφάλεια που θα δημιουργηθεί για όσους δρούν σε αυτή την αγορά και εμπλέκονται σε αυτήν. Αντίστοιχα, το θεωρώ σημαντικό από την άλλη πλευρά να δούμε τι πρέπει να ενταχθεί και τι όχι. Στις τροπολογίες μου προσπάθησα να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σαφήνειας και διαφάνειας του τι θα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο για παράδειγμα όσα για ιδιωτική χρήση ε, στοχεύουν σε ιδιωτική χρήση και όσα οδηγούν στο να υπάρξει προστασία από θερμότητα για παράδειγμα η προστασία δηλαδή που παρέχεται τι είδου είναι αντίστροφα δεν θα πρέπει τα προϊόντα τα οποία έχουν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα ή που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ε, για ιδιωτική χρήση έναντι καιρικών συνθήκων για παράδειγμα να εντάσσονται σε αυτά τα πλαίσια χρήσης. Νομίζω οι σκεψη μου είναι αρκετά σαφής και οι προθέσεις μου σαφής και στο τέλος τέλος κάπως με ενοχλούσε η διατύπωση που υπήρχε στην οδηγία αρχικά αυτό το και τα λοιπά, το ετσέτερα. Μα το ετσέτερα, το και τα είναι έκφραση νομικής αβεβαιότητας και θα προτιμούσα να μην ε, υφίσταται. Τέτοια πράγματα με κατεκτέλεση πράξης ή κατεντολήν πράξης ε, πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούν να λειτουργήσουν. Η κατεντολη πραξης πρεπει να δουμε πως μπορουν να λειτουργησουν η προταση σας μέσω των κατευθυντήριων γραμμών, προσανατολισμών, guidelines να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, ίσως θα μπορούσαμε έτσι να καθορίσουμε ποια ακριβώς άρθρα στο πεδίο εφαρμογής μπορούν να ενταχθούν και ποια όχι. Τώρα, όσον αφορά τα αντικείμενα, τα είδη για τον αθλητισμό και όσον αφορά τον συνάδελφο Βέστφαρ θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν εφόσον ο κυρίαρχος στόχος τους είναι να προστατεύεται ο καταναλωτής. Σημαντική αυτή η διαφοροποίηση. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο προανέφερα. Αν ένα τέτοιο είδος για, για αθλήματα, πώς να το πω, είναι κάτι το φθοριούχο το οποίο έχει απλά κακή ε, ας το πω έτσι, επενέργεια αλλά όχι, δεν προστατεύει πραγματικά τον καταναλωτή, τον χρήστη, ε, δεν θα πρέπει να αντάσσεται σε αυτό το πεδίο. Αντίστοιχα πρέπει να διαμορφωθεί το πεδίο εφαρμογής και ισχύω. Και είπα ότι κομμένο και αραμένο πρέπει να είναι από πλευράς πέσα ανάλογα με τις κατηγορίες κινδύνων. Και έτσι λοιπόν με τις συμβαστικές τροπολογίες θα υπάρξουν σχετικές αναφορές. Και για το δεύτερο στοιχείο πυρήνα αυτού του, αυτής ε, της πρότασης είναι η προθεσμία διάρκειας ε, και η διάρκεια πενταετίας. σε αυτή την πενταετή διάρκεια ή την υφιστάμενη αβεβαιότητα που υφίστατο να την παρακάμψω εντάσσοντας αυτά τα στοιχεία ενεργά στις διεργασίες. Είπατε αν κάτι αλλάξει τότε θα πρέπει η αρχή πιστοποίησης, ο φορέας πιστοποίησης να επανεξετάζει τα προϊόντα αυτά. Είπα με μια ε, διετή περίοδο θα μπορούσαμε να είχαμε μια λογική περίοδο διάρκειας. Όμως απορρέουν διάφορες δυνατότητες πώς θα μπορούσαμε πρακτικά να διαμορφώσουμε τα πλαίσια αυτά. Κάνατε λόγο η κυρία εισηγήτρια, για μια απλουστευμένη διαδικασία που οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προτείνουν. Μπορώ να δεχτώ εγώ ως πρόταση αυτή την απλουστευμένη διαδικασία. Τίθεται όμως ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί και πρέπει να μας προβληματίσει πώς θα το διαμορφώσουμε στην Ευρώπη. Αν ο ελεγκτικός φορέας δεν πρέπει τίποτα να εξετάσει μετά από πέντε χρόνια, αν τίποτα δεν έχει αλλάξει νομοθετικά και ο παραγωγός εξακολουθεί να παράγει τα ίδια προϊόντα, τότε θα πρέπει η αρχή πιστοποίησης να εκδίδει νέο πιστοποιητικό απαιτούνται όμως χρήματα τα οποία θα κατατίθενται για αυτό το νέο πιστοποιητικό αν όμως δεν, δεν χρειαζόταν να επανελεγχθεί τίποτα και τότε λοιπόν αν ένα επιπρόσθετο κόστος δεν θα έπρεπε να καταβάλλεται μια και τίποτα δεν αλλάζει αυτό το στοιχείο στην εκπόνηση μιας ε, συνετής λογικής λύσης, συμβαστικής λύσης πρέπει πάντα να διέπει τη δράση μας. Στην κατηγορία 1 τα προϊόντα δεν χρειάζονται ανανέωση πιστοποίησης. Γιατί δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε λοιπόν. Για την κατηγορία 2 μπορούμε να συζητήσουμε για μια αυτόματη πιστοποίηση από τον παραγωγό. Για την κατηγορία 3 για ενδεχόμενους κινδύνους θα έπρεπε να δούμε και να θυμόμαστε σε αυτές τις διεργασίες ότι στην κατηγορία 3 ετήσια διεξάγεται έλεγχος, επανεξέταση και έλεγχος αυτών των προϊόντων. Για το άρθρο 8 εδάφιο 3 προβλέπεται αυτή η ετήσια ελεγκτική δράση, αυτή η εποπτεία. Και να δούμε, σε σχέση με αυτή τη διαδικασία θα εξισώνεται με μια νέα πιστοποίηση ή όχι. Υπάρχουν παράλληλες δράσεις εδώ, παράλληλες κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθηθούν. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και να λέγαμε ότι στον τελευταίο έλεγχο, πριν δηλαδή λήξει η πιστοποίηση, να μπορεί μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης να αντικατασταθεί. Δεν θα χρειαζόντουσαν λοιπόν δύο φορές εξετάσεις, μία φορά θα εξεταζόταν και θα πλήρωνε η επιχείρηση τα τέλη αυτού του ελέγχου. Προς μια τέτοια κατεύθυνση μπορούμε να εργαστούμε για μια συμβαστική τροπολογία ώστε η εταιρεία λίγο πριν από την εκπνοή της άδεια που έχει, της πιστοποίησης που έχει, να μην χρειαστεί να ξαναπληρώνει δεύτερη πιστοποίηση. Δηλαδή να καταβάλει δύο φορές έξοδα για το ίδιο τελικά στο τέλος πιστοποιητικό. Θα μπορούσαμε να συνδυάζαμε αυτή την προσπάθεια ώστε να διαδέχεται το ένα πιστοποιητικό το άλλο και για το 209 δεσμευτικού χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι όσον αφορά τα συμπεράσματα της ε, ομάδας ε, διαχείρισης ε, ή κατευθύνσεων. Εδώ όμως δεν θα συμφωνούσα διότι θα υπονομεύαμε την νομοθετική μας προσπάθεια. Αυτή η, αυτός ο φορέας θα μπορούσε να αναλάβει νομοθετική δραστηριότητα και δεν είναι αυτό το νόημα αυτού του εγχειρήματο ενός τέτοιου φορέα δηλαδή. Και θα πρέπει εδώ να είμαστε προσεκτικοί και να επιστρέψουμε ή να παραμείνουμε σε αυτά τα οποία αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένω με αδειμονώ μάλιστα κιόλα να δω τις προτάσεις σας ποιες θα είναι ώστε να καταλήξουμε σε μια λογική αντιμετώπιση, σε μια λογική λύση αυτών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη σκέψη συγγήτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμη κυρία συγγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, χωρίς τώρα να θέλω να νοθεύσω Ε, κοιτάξτε, ίσως επειδή παίρνω νωρίτερα το λόγο από ό,τι προβλεπόταν. Εγώ δεν θέλω ε, να τα ανοθεύσω, αλλά δεν τα βλέπω και τόσο απλά τα πράγματα, γιατί έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ε, νομοθεσία. Επίσης και εγώ την τελευταία φορά είπα με απόλυτη σαφήνεια ότι τα πέντε χρόνια ισχύουν πάντα γιατί απλώς αλλάζουν τα πράγματα και νομίζω ότι απλά έπαναλαμβάνουμε λέγοντας ότι το θέμα του αμοιάντου ίσχυσε για πάρα πολλές δεκαετίες ως ε, μάλλον αμύαντος ήταν ένα πολύ καλό μέσο για την προστασία από πυρκαγιές ε, και ξέρω όμως ε, επειδή ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για να αφαιρεθεί ο αμύαντος, να μην ε, πάθουν καρκίνο τα παιδιά. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι τα 5 αυτά χρόνια θα πρέπει να παραμείνουν γιατί μόνο έτσι υπάρχει και η ασφάλεια για τις επόμενες γενιές και βεβαίως και για εμάς τους ίδιους. Θα ήθελα λοιπόν να πω και κάτι άλλο που αφορά σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ως ε, νομοθέτες ε, βεβαίως ε, και είμαστε αναγκασμένοι να δικαιολογούμεθα για, τις, για τα προγράμματά μας τα οποία και εγκρίνουμε και πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτό είναι απαραίτητο. Και εδώ ισχύει και το ίδιο. Αυτά τα οποία κάνουμε είναι απαραίτητα και μπορώ να σας πω με απόλυτη έννοια ναι, είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητο όσον αφορά αυτές, αυτούς τους εξοπλισμούς προστασίας να υπάρξουν κάποιες διορθώσεις. Είναι απαραίτητες αυτές για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Έτσι λοιπόν, εάν για ε, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς λόγους ε, χρησιμοποιούνται αυτοί οι εξοπλισμοί, πρέπει όσοι χρησιμοποιούν αυτούς τους εξοπλισμούς να έχουν το κατάλληλο υλικό, αλλά επίσης ε, να μπορούν και να είναι σίγουροι ότι προστατεύεται η ζωή τους. Όλα αυτά λοιπόν ε, θέλω να σας τα παρουσιάσω με ένα εύλογο παράδειγμα, ένα παράδειγμα το οποίο αφορά όλους μας, το οποίο μπορεί να μας αφορά όλους μας. Αναφέρομαι ε, στους πυροσβέστες που τους χρειαζόμαστε ε, παντού και οι άνθρωποι οι οποίοι κατ' ουσίαν ε, χρησιμοποιούν τη ζωή τους ε, για να βοηθήσουν άλλους, αυτοί βεβαίως θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι απολαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή σημασία για τη ζωή τους έτσι ώστε ε, να χρησιμοποιούν τη ζωή τους για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Ε, και πρέπει να ξέρετε τι, ξέρω τι λέω, γιατί ο άνδρας μου είναι γιατρός και αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να περάσει αυτός ο κανισμός. Η διαφορά ανάμεσα σε εμάς, ε, κυρία εισηγήτρια και την δική μου την πολιτική ομάδα είναι ότι εμείς ή εσείς ακολουθείτε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εσείς προτείνετε να μειωθούν κάποιοι τομείς εφαρμογής παραδείγματο χάρη τι επιτόπιε έρευνε, τι βρίσκεται πολύ σημαντικέ και θα, ήθελα, θα θέλετε να υπάρχει και μια ε, δήλωση συμμόρφωση τα πέντε χρόνια, τα επέκνα ήδη την τελευταία φορά και το κάνω και σήμερα. Εγώ αντίθετα θεωρώ την πρόταση της Κομισιόν, την θεωρώ καλή. Βεβαίως και χρειάζεται διορθώσεις μόνο προς διαφορετική κατεύθυνση, προς τα εκεί που προτείνω εγώ. Τώρα, όσον αφορά την πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αφενός ε, τους κατασκευαστές οι οποίοι ε, πρέπει να ε, δείχνουν κάποια εμπιστοσύνη σε αυτά που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει το ΠΕΣΑ θα πρέπει να αναφέρεται και ως ΠΕΣΑ αυτή λοιπόν η εμπιστοσύνη αυτή την εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να την αφήσουμε μόνο στα χέρια των οικονομικών παραγόντων. Εγώ είμαι πολύ ε, σοσιαλίστρια για να δω κάτι διαφορετικό. Πρέπει τους ε, κρατικούς ε, φορείς να τους ενισχύσουμε και αυτή η, ο έλεγχος αγοράς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και καλός και να λάβει χώρα το στομότερο δυνατόν. Για να γίνουν όλα αυτά είναι απαραίτητο να υπάρχει χρόνος και δηλώσει συμβατότητα ε, που θα επικρέμανται σε ένα προϊόν. Βεβαίω και θέλουμε να πλουστεύσουμε την κατάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η γραφειοκρατική επιβάρυνση είναι ελάχιστη, όμως η ασφάλεια που προκύπτει πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν λέω για άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Εγώ την πρόταση της Κομισιόν με όλες τις τροπολογίες που έχω καταθέσει την βρίσκω πολύ καλά ε, και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω τελικά τι θα γίνει με τις συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, ευχαριστώ πολύ. Μου δείτε ή δείτε μάλλον να πει το κύριο Ροσφό. Ναι, καταρχά ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του Ρόμπερτ που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρου του την εισηγήτρια για το έργο τη πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Ρόμπερτ ε, ήδη έχει εκφράσει τι απόψει του για αυτό το ζήτημα και εδώ αλλά και στη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να συνοψίσω κάποια βασικά για αυτόν σημεία αλλά και για την ομάδα μας σημαντικά σημεία. Η δική μας πολιτική ομάδα στηρίζει τις ισχυρές ε, απαιτήσεις για αυτό τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ε, γιατί η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, βέβαια, στηρίζουμε και την εναρμόνιση της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρχικό σύστημα ήταν ικανοποιητικό, άρα στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια τομή και να αλλάξουμε άρδιν το ρυθμιστικό πλαίσιο. Απλά με αυτή την πρόταση έχουμε την δυνατότητα να βελτιώσουμε, να εξυγχρονίσουμε, να απλουστεύσουμε και να διευκρινίσουμε. Χαιρετίζουμε τη δουλειά της Προέδρου μας και η συγγήτρια στην προκειμένη περίπτωση. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού στο PPE, ε, δηλαδή ε, στα ατομικά μέσα προστασίας ε, κατά της ε, θερμότητας, ε, της υγρασίας. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη και το διοικητικό άχθος και η σχέση που έχει και η αναλογία που έχει με τη μείωση των κινδύνων. Δηλαδή, όχι κάποιες, κάποια μελιτέοι κίνδυνοι να καλύπτονται, Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες σε σχέση με τα σημεία αυτά για τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την δήλωση συμμόρφωσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κανονισμού ότι δηλαδή γνωρίζουμε ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσει του κανονισμού το προϊόν. Οι οικονομικοί παράγοντες θα πρέπει να έχουν την επιλογή είτε να δίνουν ε, ένα αντίγραφο υλικό είτε ένα σύνδεσμο στο διαδίκτυο όπου θα μπορεί ο καταναλωτή να πάρει αυτέ τι πληροφορίε. Ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση των προϊόντων, ξέρουμε ότι οι καταναλωτέ, οι χρήστε ε, το χρειάζονται αυτό. Θα πρέπει λοιπόν οι οδηγίε χρήση να περιλαμβάνουν τι σχετικέ διατάξει. Οι αρχέ εποπτεία τη αγορά θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση όπως και οι καταναλωτές ε, και οι χρήστες, είτε σε έντυπη μορφή είτε στο διαδίκτυο και οι οδηγίες προς το χρήστη θα πρέπει να είναι ευλήπτες, να επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα, όπως επίσης εύκολα προσβάσιμο θα πρέπει να είναι και το πιστοποιητικό συμμόρφωση από τις αρχές εποπτές της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τώρα την εισαγωγή ή μη εισαγωγή, η θέσπιση μιας επιχρεωτικής ε, περίοδου ισχύω για τα πιστοποιητικά Κάποιοι θα ήθελαν οποιαδήποτε αναφορά σε ένα μέγιστο ε, διάστημα ισχύω ε, για αυτό το πιστοποιητικό εξέταση που βλέπετε τη πρόταση τη Επιτροπή να μην ισχύει, ενώ άλλοι θα ήθελαν να επεκταθεί, να επιμηκυνθεί σε 10 χρόνια. Αυτό να είναι το ελάχιστο διάστημα. Και άλλοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα μέσα προστασία. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε από κοινού. Πιστεύω, όπως και η Κομισιόν και οι άλλοι προείπαν, ότι θα πρέπει να ορίσουμε την ε, περίοδο ισχύω και θα πρέπει να μπορούμε να επιτρέπουμε ε, την ε, περιοδική εξέταση της έγκρισης τύπου κατά γενικό κανόνα. Επίσης θα πρέπει να είναι απλουστευμένη η διαδικασία για την ανανέωση των πιστοποιητικών όταν βέβαια δεν απαιτούνται ξεκάθαρα επιπλέον έλεγχοι, αν δεν έχει αλλάξει το προϊόν, αν δεν έχουν αλλάξει τα πρότυπα και όταν το προϊόν εξακολουθεί να πληρεί τις ε, βασικές απαιτήσει, ε, υγείας και ασφάλεια. Φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τον καλύτερο προσδιορισμό των όρων και προποθέσεων αυτών. Πρώτη στη σημασία όμω έχει να οριστούν ξεκάθαρα περιπτώσεις όπου αυτή η απλουστευμένη διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και έτσι να έχουμε σχεδόν αυτόματη επαναπιστοποίηση. Στηρίζουμε επίσης τις τροπολογίες 160 και 238 που έχουμε θα σας με την εισηγήτρια. Δεν στηρίζουμε τις τροπολογίες 157, 234, 235, 236 και 237. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε καλή συνεργασία και θα συνεργαστούμε και με τους κοιόδους και με την εισηγήτρια και στη συνέχεια. Αυτά είναι τα λόγια του Ρόμπερτ που σας χαιρετά. Thank you. Um, at this stage... Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Στρέφομαι στους άλλους κοιόδης. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κανένας άλλος κοιόδης εισηγητής. Θα έδινα τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και τις τροπολογίες και για το ότι μας δίνετε τον λόγο να παρέμουμε. Στην τελευταία συνεδρίαση και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να ε, λέμε ότι υποστηρίζουμε την άρση της εξαίρεσης ε, όσον αφορά τα, τις συσκευές αυτές ε, που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Είχαμε πει και κατά την τελευταία συνεδρίαση ότι θα υποστηρίξουμε μια συμβαστική λύση που θα είναι αποδεκτή από τον συνομοθέτη. Όμως, τούτων λεχθέντων θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι, διότι η τροπολογία 247 και 173 τι προτείνουν. Προτείνουν να εξαιρεθεί από το εύρος, να εξαιρεθούν προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο εύρος στο πλαίσιο της υφιστάμενης οδηγίας. Το συμβαίνει με την τροπολογία 273 όσον αφορά καθαριστικό υλικό για παράδειγμα ή δράση καθαριστική που βρίσκεται στο ε, εύρος της ε, υφιστάμενης οδηγίας και σε σχέση με την τροπολογία επίσης 147 όλα τα προϊόντα για ιδιωτική χρήση που δεν συνδέονται με κίνδυνο ζωής κάλυψη κινδύνου, προστασία από κίνδυνο ζωής Δηλαδή εξαιρούνται για παράδειγμα γυαλιά ηλίου και τα λοιπά ως ε, ξεχωριστή κατηγορία. Επίσης έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την αναφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα στα άρθρα, στα επιμέρους άρθρα. Συμβαίνει αυτό σε σχέση με τις τροπολογίες 269-262. Θα ήθελα να σας πω ότι το πρόβλημά μας αφορά την υλοποίηση της νομοθεσίας στην πρακτική εφαρμογή, διότι πολύ συχνά χρειάζεται, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήσεις Δηλαδή ποια είναι η πρόθεση του νομοθέτη για να, αναφέρεται, να αναφέρονται συγκεκριμένα προϊόντα και τι γίνεται με τα υπόλοιπα, εντάσσονται ή όχι στις διατάξεις αυτές. Τώρα, όπως προτείνεται σε σχέση με την τροπολογία 154 και την 182, αυτές οι διατάξεις θεωρούμε εμείς μπορεί να εξεταστούν στην νομοθεσία για την διάταξη και τις, ε, ε, για τις διατάξεις όρων εργασίας. Δεν βρίσκεται όμως στο πλαίσιο αυτό, δεν βρίσκονται στο πλαίσιο αυτό για την ασφάλεια δηλαδή. Εδώ γίνεται λόγος για εργονομικά θέματα που αφορούν θέματα ε, συνθήκων εργασίας και όχι στο πλαίσιο ασφάλειας. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες 237 όσον αφορά τον καθορισμό της ε, χρονικής διάρκειας θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι εκείνοι οι οποίοι επικαιροποιούν τα προϊόντα τους ώστε να είναι το τα τελειότερα δυνατά <clears throat> βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με εκείνους που λένε ότι έχουν διαβίου ε, πιστοποιητικό το οποίο ισχύει διαβίου σε σχέση με τις ε, ε, υπόλοιπες τροπολογίες, το πρόβλημα το οποίο ε, δημιουργείται είναι ότι το πιστοποιητικό μπορεί να συνεχίσει να ισχύει μετά την απόσυρση του εναρμονισμένου, των εναρμονισμένων στοιχείων. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αν έχουμε εδώ ταυτοποίηση κινδύνου ζωής, τότε αυτές οι διατάξεις θα επέτρεπαν η πιστοποίηση να συνεχίσει να ισχύει και να έχει ισχύ. Τώρα, εδώ το πρόβλημα πάντα αναφύεται ποιος είναι ο λόγος να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή. Αν υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την ε, ανθρώπινη ζωή δημιουργείται ένα νέο διαφορετικό καθεστώς. Σε σχέση με αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται εδώ σε ένα άρθρο τομεακού χαρακτήρα νομοθετικά είναι μείζον πρόβλημα. Και αυτό γιατί, διότι η ουσιαστικές απαιτήσει αφαιρούν τον τομέα ασφάλειας. Αυτό που κάνει η τομεακή ε, ρύθμιση είναι να καθοριστούν οι διατάξεις που πρέπει σύμφωνα με αυτές να συμμορφώνεται ο παραγωγός, η εταιρεία που παράγει αυτά τα προϊόντα. Αν υπάρχουν κίνδυνοι θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να γίνει προσπάθεια συμμόρφωσης Σήμερα για μια γενική αναφορά όσον αφορά για παράδειγμα τον συνομοθέτη δεν χρειάζεται να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένων διατάξεων. Και πάλι όμως σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων διεξάγονται αυτές οι συζητήσεις. Αν λοιπόν συμπεριλαμβάνεται αυτό το άρθρο τότε υπάρχει επιθυμία να ισχύουν αυτοί οι κανόνες και να εφαρμόζονται. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα για μας που δημιουργούνται σε σχέση με τη λειτουργία Όλες οι διατάξεις για την ασφάλεια πρέπει μέσα στο πλαίσιο των νομοθετικών να εντάσσονται και να λειτουργούν. Καλωσορίζουμε τις τροπολογίες 106 και 138 που ε, καθορίζουν τα θέματα των ε, εξετάσεων αν τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με ένα προϊόν. Όσον αφορά τροπολογίες ε, σε σχέση με την αντανάκλαση ε, φθορείου είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα το οποίο το έχουμε πολλές φορές συζητήσει να δούμε πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να διευθετηθεί. Εμείς θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι καλό θα ήταν αν θα μπορούσαμε να είχαμε αντικειμενικά κριτήρια. Η τροπολογία 277 για παράδειγμα καθορίζει κάποια κριτήρια τα οποία θεωρούμε ότι θα άξιζε να εξεταστούν γιατί είναι καλύτερο να υπάρχει αναφορά σε αντικειμενικά κριτήρια παρά να αναφερόμαστε σε κάποια γενικόλογα που θα έχριζαν ερμηνείας ε, άρθρα ή σκεπτικά. Και με βάση αυτό θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αντικειμενικά κριτήρια. Για την τροπολογία 190 θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ε, θέμα των, των εικόνων, των συμ, ε, Επίσης τώρα σε σχέση με την υποχρεωτική πιστοποίηση 112 για παράδειγμα τροπολογία και άλλες συναφείς είναι ένα θέμα το οποίο είχε συζητηθεί όταν είχε διεξαχθεί η αρχική συζήτηση για συνεννόηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Τότε η συμφωνία που είχε ε, προσεγγιστεί ήταν ότι δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα αυτή η πιστοποίηση. Υπήρξαν όμως είχαν κάποια προβλήματα και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνει η προσπάθεια να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε την συμφωνία εκείνη που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά το παρελθόν. Κατανοούμε ότι μπορεί αυτό να αποτελεί μια δυνατότητα για το μέλλον, μια τέτοια υποχρεωτική πιστοποίηση. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ, εισηγείτε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τα σχόλια. Θα είναι σαφές αυτό που ε, φυσικά και χρειαζόμαστε σαφήνεια σε ό,τι αυτό το εφαρμογή να ευχαριστήσω την Κομισιόν και για αυτό που είπε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προτιθέμεθα την ασφάλεια του εξοπλισμού παραδείγματος χάρη που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες ε, να την ε, υποβαθμίσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν καταθέτουμε τροπολογίες που υποβαθμίζουν την ασφάλεια, επαγγελματικού εξοπλισμού ασφάλεια. Σίγουρα θα καταθέσουμε τροπολογίες. Η λέξη και λοιπά και το etc. Ε, είναι στο φάκελο που χρησιμοποιείται εδώ και 25 χρόνια, αλλά ίσως στη σύγχρονη γλώσσα θα μπορούσε πράγματι να απαντήσει σε μία ε, σκέψη, αλλά όχι στο σώμα του κειμένου. Θα βρούμε κάποια αναλλακτική διατύπωση. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα αφαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής ο προσβεστικός εξοπλισμός. Δεν ξέρω γιατί ε, τέθη αυτό το θέμα. Τα πέντε χρόνια Ήθελα να ακούσω τις απόψεις ε, των συναδέλφων. Εγώ πάντα είχα σαφή άποψη. Είχα συνυπογράψει και τροπολή με τον κύριο Ροσφόρ, η οποία λέει ότι αν ένα ε, πιστοποιητικό σε ισχύ ε, κοντεύει να λήξει και υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, μάλλον και δεν υπάρχουν σημαντικέ αλλαγέ, δεν χρειάζεται οι μικρέ εταιρείε τουλάχιστον να περάσουν από πολύ δυσκίνητε γραφειοκρατικέ διαδικασίε για την επανέκδοση πιστοποιητικού. Νομίζω ότι το ίδιο λέει και η Κομισιόν. Μας έχει βοηθήσει στη διατύπωση και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι επ' αυτού. Και βέβαια για ένα πολύ συγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ε, Ασφάλειας για την αποστευμένη διαδικασία κάποιοι κλάδοι όπου δεν υπάρχει ε, μια καταληκτική μία αυτόματη. Τι γίνεται εκεί, ε, τέθη αυτό το θέμα από κάποιους ε, ενδιαφερομένους. Δεν έχουμε όμως την πρόθεση να αφήσουμε να νοηθεί ότι οι φυστάμενες διαδικασίες ανανέωσης ή ετήσιοι έλεγχοι που ανέφερε ο Σκιώδης από το ΕΛΚ δεν θέλουμε να αφαιρεθούν αυτά, δεν θέλουμε να καταργηθούν, απλά πρέπει να βρούμε μία λύση που να μπορεί να λειτουργήσει για προϊόντα που δεν έχουν μια καταληκτική μερομηνία ισχύω πρώτον και δεύτερον όταν δεν έχουμε σημαντική αλλαγή στην νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά μίλησε για την τροπολογία αυτή που λέει αν ένα πρότυπο έχει αποσυρθεί, τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Αν λοιπόν έχει αποσυρθεί ένα πρότυπο γιατί είναι το προϊόν επικίνδυνο για τη ζωή είναι άλλο από το αν ε, υπάρχει απλά μια επικαιροποιημένη μορφή του ή αντικατάσταση. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να καταλήξουμε σε μια περίοδο όπου δεν θα υπάρχει κανένα εξοπλισμός ασφαλείας, ούτε ο παλιός το καινούριος. Άρα στη μεταβατική, πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική φάση μεταξύ του παλαιότερου και του νεότερου προϊόντος για να μπορούν να προμηθευτούν τον εξοπλισμό ασφαλείας. Εργαζόμενοι Επίση. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν τα γυαλιά ηλίου. Ό,τι είναι μέσα, δηλαδή στο οποίο εφαρμογή πρέπει να παραμείνει. Επιτόπι έλεγχη. Ναι, πράγματι πρέπει να είναι σαφείς οι τροπολογίες. Θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα δεύτερο γύρο, ίσως αυτό. Μην υποτιμάτε παρακαλώ τη σημασία του να έχουμε εργονομικό εξοπλισμό. Παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση την ε, Διεθνή Μέρα της Γυναίκας ε, για εξοπλισμό ασφαλείας ε, κατάλληλο για γυναίκες στον τομέα της μηχανικής, της επιστήμης. Αν δεν προσαρμόζεται και δεν σε προστατεύει ο οργανισμός, ο εξοπλισμός ε, δεν είναι καλά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να μπορούν να βρουν εξοπλισμό τον οποίο, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και ότι είπατε για την αρχή της προφύλαξης μας βρίσκει σύμφωνους. Για τον αθλητικό εξοπλισμό ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμό μεταξύ μας. Καταλαβαίνω τι λέει η Κομισιόν για τη χρήση της λέξης fashion. Ίσως από νομικής πλευράς αυτό, η μόδα, ο σειρμός, να είναι δύσκολο να οριθεί. Τι Θα δούμε όμως. 78-209 θα τις δω αυτές τις τροπολογίες. Για τη δήλωση συμμόρφωσης. Η συμμόρφωση πρέπει να διατίθεται σε έντυπη μορφή ή επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Ναι, νομίζω εγώ. Οι χρήστες πρέπει να έχουν σαφείς οδηγίες. Άλλο είναι αυτό από το πώς διατίθεται το πιστοποιητικό ή η δήλωση Ο διανομέας, ο κατασκευαστής, άλλο είναι να έχει αυτή τη δήλωση μόρφωσης και άλλο οι καταναλωτές, οι χρήστες να έχουν οδηγίες χρήσης. Ίσως δεν έγινε αντιληπτό ακριβώς αυτό που εννοούσα ή αυτό που εννοούσατε εσείς, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουν σαφείς οδηγίες οι χρήστες. Και χαίρομαι που η Κομισιόν συμφωνεί με τα σχόλια που έκανα για αυτά τα εικονογράμματα, τα pictograms που είναι κάποιες φορές παραπλανητικά ή καθόλου σαφή. Αυτά είναι τα βασικά σημεία Προς το παρόν έχω συντάξει κάποιες τροπολογίες συμβιβαστικέ, σχέδιο είναι ακόμη και ελπίζω να τις δεχθούν περισσότεροι συνάδελφοι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Εξέταση συμβαστικών τροπολογιών στην Επιτροπή μας στις 20 Απριλίου και ψηφίζουμε στις 23 Απριλίου στην Επιτροπή μας και εντολή έθραξης διαπραγματεύσεων ελπίζουμε να είναι για το Μάιο του 2015. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια, ευχαριστούμε τους σκιώδεις και σας δίνω τη σκητάλη, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε την απόψινή συνεδρίαση. not any other business... Για τα διάφορα δεν ξέρω αν έχετε κάτι. Τελειώσαμε. Thank you. the next date... Επόμενη ημερομηνία 20 Απριλίου στις 3 τα απόγευμα.